Συνάδελφοι από τα Εθνικά Κοινοβούλια, αγαπητοί συνάδελφοι από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σας παρακαλώ να καθίστε. Θα αρχίσουμε σε λίγα δευτερόλεπτα τη συνεδρίασή μας και χαίρομαι που σας βλέπω όλους εδώ. Πρόκειται για ένα θέμα πάρα πολύ σημαντικό Νομίζω ότι είναι προσφυλές ε, το θέμα αυτό για μένα ως ε, μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επί πέντε χρόνια. Ήμουνα τακτικό μέλος, όχι το πρόεδρος, ο κύριος Ρόλ που κάθεται δίπλα μου. Και ήταν μια δραστηριότητα πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, οφείλω να σας ομολογήσω, διότι η ενέργεια είναι νομίζω το ε, σημαντικότερο θέμα για τους περισσότερους από τους πολίτες μας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κοινή αγροτική πολιτική. Δεν έχουμε καμιά, κανένα πρόβλημα με την διατροφή, με τα τρόφιμα. Και ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι σε πάρα πολλά μέρη του κόσμου είναι ε, το σημαντικότερη δυσκολία το, τα τρόφιμα και το είδωρ, το νερό. Το πρόβλημά μας ε, είναι ο εφοδιασμός ο ενεργειακός. Συνεπώς, έχουμε να κάνουμε με σημαντικότατο θέμα σήμερα και το αντιμετωπίζουμε με μεγάλη σοβαρότητα διότι είναι πρόκληση και ακόμα και απειλή για τους πολίτες μας. Ας το θέσουμε έτσι. Θα ήθελα ε, τώρα να περάσω στη μητρική μου γλώσσα όπως γίνεται στην Επιτροπή Ήτρε εφόσον θα χρησιμοποιήσουμε τις δεξιότητες και τις γνώσεις των διερμηνέων μας. Πορτογαλικά. Υπουργέ Κόβατς, αξιότιμοι συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι βουλευτές. Θα ήθελα να σας καλωσορίσω και πάλι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα μιλήσω στη μητρική μου γλώσσα για ένα ζήτημα που είναι κέριο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, το θέμα της ενέργειας. Δεν υφίσταται οικονομική ανάπτυξη αν δεν σημειώσουμε πρόοδο ως προς τον ενεργειακό ανεφοδιασμό. Σε αυτήν την ε, μεικτή συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των Εθνικών Κοινοβουλίων που συνιστά πλέον παράδοση βάσει της συνθήκης της Λισαβόνας γιατί γνωρίζετε πως έχουν νέα δικαιώματα πλέον τα Εθνικά Κοινοβούλια δυνάμει της συνθήκης αυτής και δύνανται να επηρεάσουν την εξέλιξη της νομοθεσίας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ας επιστρέψουμε τώρα στο σημερινό μας θέμα. Ε, μεταξύ των στόχων είναι και η τόνωση της ανταγωνιστικότητας, η χρήση των εφιών ενεργειακών συστημάτων και η ανάπτυξη ενεργειακών υποδομών. Δηλαδή, με άλλα λόγια, ο στόχος είναι να οικοδομήσουμε μία εσωτερική ενιαία αγορά ενέργειας όπου θα ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα διότι ενίοτε υπάρχουν εθνικά μονοπόλια όπως όλοι γνωρίζουμε αλλά όχι στην εσωτερική αγορά. Τι σημαίνει η ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά. Σημαίνει ότι χρειαζόμαστε υψηλότατες επενδύσεις για να εξασφαλίσουμε τη διασύνδεσιμότητα των εθνικών μας δικτύων και για να εγκαθιδρύσουμε ευφυή ενεργειακά συστήματα. Χρειάζεται λοιπόν πέρα από τι επενδύσει και έρευνα. Έρευνα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ούτω ώστε να μπορέσουμε να αναβαθμίσουμε τα τεχνολογικά συστήματα που χρησιμοποιούμε για τον ενεργειακό ανεφοδιασμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Πριν από ένα χρόνο περίπου, προτάθηκε η δημιουργία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ενέργειας. Δεν επιθυμούμε να αλλοιωθεί αυτός ο στόχος. Το αντίθετο, ε, επιθυμούμε την συγκρότηση ενός ενιαίου πλαισίου όπου θα εγγράφονται όλες οι δράσεις που σχετίζονται με τον ενεργειακό εφοδιασμό. Ακόμη και το θέμα της ενεργειακής αλληλεγγύης ε, στην Ένωση, διότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση η εξάρτησή μας είναι της τάξης του 55% για τον ανεφοδιασμό από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ευχερέστερο να διαπραγματευόμαστε λοιπόν συμβόλαια και συμβάσεις ανεφοδιασμού σε εσωτερικό επίπεδο. Αν καταλήξουμε σε συνένεση βέβαια σε ένωση. Εάν καταλήξουμε στα πλαίσια αυτών των διαπραγματεύσεων σε μια ενιαία θέση θα είναι και πιο κρατεά και έτσι θα δημιουργήσουμε μια πιο ανταγωνιστική, μια ενισχυμένη ενεργειακή αγορά με αποτέλεσμα την περικοπή του κόστους, ε, πράγμα ενδιαφέρον φυσικά και για τους παραγωγούς αλλά και για τους καταναλωτές. Πρέπει να διευκολύνουμε την έρευνα, να προστατεύσουμε με τις νέες τεχνολογίες ε, το περιβάλλον. Αυτό θα καταστήσει εφικτό μόνο αν συνεργαστούμε. Περί αυτού πρόκειται όταν μιλάμε για την ενεργειακή ε, κοινότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να συνεργαστούν για να συγκροτηθεί ένα ειδικό, ενιαίο πλαίσιο για αυτήν την ενεργειακή αγορά. Δεν πρόκειται για ε, ίδρυση νέων θεσμών ή εισαγωγή τροπολογιών ε, στη συνθήκη. Όχι. Ο στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε ένα κίνητρο, ούτω ώστε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης να συμπορευτούμε ε, για τα ενεργειακά ζητήματα, για τα μεγάλα προγράμματα πράγματα τώρα, δηλαδή για τους ενεργειακούς ε, διαδρόμους ε, σε μακροκλίμακα ή οποιαδήποτε άλλα προγράμματα ε, που τοποθετούνται στην μικροκλίμακα Παραδείγματο χάρη τα ενεργειακά δικτύα, γιατί μην ξεχνάτε την πρόσφατη κρίση που βιώσαμε για το φυσικό αέριο. Λοιπόν, το δίδαγμα που αντλούμε είναι ότι απαιτείται ενεργειακή αλληλεγγύη και συνεργασία σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα συγχαρητήρια προ τον Πρωθυπουργό Όρμπαν που ανέπτυξε το πρόγραμμα τη ενεργειακή γέφυρα ανάμεσα στη Βαλτική ε, θάλασσα και τον Εύξηνο Πόντο. Ε, διασύνδεση για τη μεταφορά φυσικού αερίου. Ε, τώρα, ως προς ε, τα προγράμματα που αναπτύχθηκαν ε, πριν από χρόνια όταν εγώ ήμουν Πρωθυπουργό και το ίδιο και ο κύριος Όρμπαν εξάλλου αυτή η γέφυρα ε, κατέδειξε τη σημασία της. Σας παραπέμπω ας πούμε στον αγωγό Ναμπούκο. Ήταν η πρώτη ε, ενεργειακή διασύνδεση για την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση σε μικροκλίμακα τώρα στις πόλεις. Θα πρέπει να τροποποιήσουμε τα απερχαιωμένα συστήματα θέρμανσης, ε, δηλαδή να χρησιμοποιούμε τα ηλιακά πάνελ, την ολική ενέργεια, να εφεύρουμε νέες ενιαίες λύσεις για την Ευρωπαϊκή Ένωση για να διασυνδεθούν τα εθνικά μας συστήματα. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, έχουμε συστήσει μία διακομματική ε, ε, ομάδα με τίτλο Urban που έχει επιληφθεί αυτού του ζητήματος της αστικής θέρμανσης. Τέλος, θα ήθελα να ζητήσω από τους συναδέλφους, όταν έρχεστε σε επαφή ε, με τους πρόεδρους των Εθνικών Κοινοβουλίων ή με τα μέλη της κυβέρνησης της χώρας σας, ε, να ε, τονίζετε αυτά τα ενεργειακά ζητήματα, να τα συζητήσετε μαζί τους και να έχετε υπόψη σας αυτήν την ευρωπαϊκή διάσταση που προανέφερα, γιατί έτσι θα είναι πολύ πιο εύκολο να προστατεύσουμε το περιβάλλον και να καταστήσουμε ε, πιο ασφαλή τον ενεργειακό αναφοδιασμό ε, στο χαμηλότερο δυνατό κόστος. Γνωρίζουμε ότι οι τιμές ποτέ δεν θα είναι χαμηλές, αλλά ο στόχος είναι να είναι οι τιμές προσιτές, ούτως ώστε να είναι και ανταγωνιστικοί. η οικονομία μας. Θα ήθελα να σε υπενθυμίσω ε, ότι διοχετεύτηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 4 ευρώ και θα έπρεπε η επένδυση αυτή να μας οδηγήσει σε αυτά αποτελέσματα Δηλαδή, Θα θέλαμε να υπάρξουν νέες συγκεκριμένες δράσεις, ξεκινώντας από τα πρώτα 22 εκατομμύρια επενδύσεων που πρέπει να γίνουν και ε, θα ήθελα να τονίσω επίσης ε, τη σημασία που έχουν αυτές οι δράσεις στα πλαίσια της δημιουργίας της ενιαίας ε, αγοράς. Τώρα, για τον προπολογισμό της Ένωσης μετά το 2013 θα πρέπει να προσδώσουμε την, ε, το δέον ειδικό βάρος, αν θέλετε, στο θέμα της ε, ενέργειας, ε, την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών. Θα ήθελα να τονίσω ότι το θέμα της χρηματοδότησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχει ιδιαίτερη σημασία κυρίως στις διαπραγματεύσεις που έχουμε με την Επιτροπή και το Συμβούλιο. Μην ξεχνάτε τις προσδοκίες των πολιτών ε, της Ένωσης. Πάντως, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα Εθνικά Κοινοβούλια ασχολούνται επισταμένα με τα ενεργειακά ζητήματα και σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και σε ε, εθνικό επίπεδο, σε κάθε μεμονωμένο κράτος μέλο ε, διότι ουδής μπορεί να απομονωθεί ενεργειακά ε, στην γυραιά Ήπειρο. Χρειαζόμαστε ε, και οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι εξακολουθούν να υφίστανται αυτές οι ενεργειακές νήσοι μέσα ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα πρέπει να έρουμε αυτούς τους φραγμούς για να λειτουργεί πιο εύρυθμα το σύστημα και να βασίζεται στην ενεργειακή αλληλεγγύη. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ευχαριστώ που θα συμμετάσχετε σε αυτή την τόσο σημαντική συζήτηση. Κύριε Πρόεδρε Μπούζεκ, εξ ονόματος όλων των συναδέλφων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των Εθνικών Κοινοβουλίων θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα που συγκαλέσατε αυτή τη διάσκεψη εδώ στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα Σας ευχαριστώ επίσης για την παρουσία σας διότι έχετε τόσα άλλα καθήκοντα και χαιρόμαστε που είσαστε εδώ παρόν και αυτό δείχνει στους καλεσμένους μας από τα Εθνικά Κοινοβούλια ότι αυτή η συνεργασία με τα Εθνικά Κοινοβούλια σας ενδιαφέρει ιδιαίτερα και ότι το θέμα της ενέργειας είναι ένα θέμα στο οποίο αποδίδεται ιδιαίτερη προτεραιότητα. Σας ευχαριστώ που ήρθατε εδώ και που μας δώσατε την δυνατότητα να έρθουμε σε επαφή με τους συναδέλφους και να γενιάσουμε την διάσκεψη αυτή της Επιτροπής Ήτρε. Χαιρετίζω όλους τους συναδέλφους των Εθνικών Κοινοβουλίων και κυρίως τον κύριο Πάλκοβατς ο οποίος είναι ο Υφυπουργός Ενέργειας στην Ουγγαρία η, την Προεδρία, η Προεδρία η οποία αντιπροσωπεύεται αρκετά ο Herbert Ρουλ είναι παρόν. Ο Ρουλ, ο, ο ε, Γενικός Διευθυντής Ενέργειας, ο οποίος εκπροσωπεί τον ε, Επίτροπο Oettinger, ο οποίος δεν μπόρεσε να έρθει. Ο κύριος Λόβ τον, τον εκπροσωπεί και χαιρετίζω επίσης ε, τον Αντάλ Ρογκάν, ο οποίο είναι πρόεδρο τη Επιτροπή Οικονομικών Θεμάτων Τεχνολογία Πληροφορικής της Πληροφορίας του Κοινοβουλίου τη Ουγγαρία, και θα ήθελα τώρα να δώσω τον λόγο πρώτα απ' όλα στον κύριο Ρογκάν, διότι θα προεδρεύσουμε ε, μαζί αυτήν τη συνεδρίαση. Σα δίνω τον λόγο κύριε Ρογκάν. Én is nagyon χαίρομαι και εγώ που σήμερα υπό ουγγρική Προεδρία θα έχουμε την ευκαιρία να πραγματευτούμε αυτό το τόσο σημαντικό ζήτημα. Για μας είναι ιδιαίτερα κέριο και το έχουμε αναδείξει προτεραιότητα τη Προεδρία μα. Χαιρόμαστε ιδιαίτερω ε, που δεν έχει εγγραφεί αυτό το σημείο σε ένα απλό σημείο της μίσιας διάταξης, αλλά συνδυάζεται με άλλα ζητήματα που έχει σημειωθεί πρόοδος. Ε, πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλήξουμε τελικά σε κάποια συνένεση για κάποια βασικά ζητήματα όπως τη δημιουργία μιας κοινή αγοράς για το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο μέχρι το 2014 και πιστεύω πως θα ήταν σκόπιμο να κάνουμε έναν απολογισμό της βασικότερης πρόοδου που έχει σημειωθεί στον τομέα αυτό και να διερευνήσουμε ε, τους τρόπους χρηματοδότησης των νέων ενεργειακών υποδομών που απαιτούνται, καθώς και να εξετάσουμε το θέμα της χρηματοδότησης των μεγάλων ενεργειακών προγραμμάτων. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας δώσατε την ευκαιρία να συμμετάσχουμε στη σημερινή συνεδρίαση. Ευχαριστώ εκ των προτέρων όλους τους παρισταμένους για την παρουσία, της, ε, παρουσία τους εδώ σήμερα και θα προσθέσω στη συνέχεια και ε, άλλα ε, στοιχεία σε μελλοντικές παρεμβάσεις μου δηλαδή. Ο κύριος Ρόιλ. Λοιπόν, ας αρχίσουμε τώρα με την μερίσια διάταξη. Θα πρέπει να είμαστε λίγο αυστηροί με το χρόνο για να προλάβουν όλοι να παρέμβουν. Στρέφω προς το Γενικό Διευθυντή ε, για τα ενεργειακά ζητήματα, Φιλίπ που αντικαθιστά τον Επίτροπο Έτιγκερ. Έχετε το λόγο. Uh, Ευχαριστώ πολύ για αυτήν ε, την πρόσκληση σε αυτήν την σημαντικότατη συζήτηση μεταξύ των μέλη του Κοινοβουλίου του Ευρωπαϊκού και των Εθνικών Κοινοβουλίων. Η ευρωπαϊκή πολιτική ε, είναι μια επικοδομητική ε, οργάνωση μεταξύ εθνικών συζητήσεων στις Εθνικές Βουλές και κοινοβουλευτικών συζητήσεων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ε, πρόκειται για την συνειδητοποίηση της εξάρτησης που έχουμε από τις ενεργειακές πηγές. Πρέπει να αναπτύξουμε ανταγωνιστικές πηγές ενέργειας, διαφορετικές, ούτως ώστε να είμαστε αυτόνομοι και να έχουμε ε, ανταγωνιστικότητα στο ενεργειακό επίπεδο και στις τιμές της ενέργειας. Έχουμε οπωσδήποτε αναλάβει ένα έργο μακρόπνο. Θέλουμε να ε, θεσπίσουμε ένα οικονομικό σύστημα ως προς την ενέργεια που να ε, μην έχει πολύ υψηλέ τιμές και να μην βλάπτει το περιβάλλον. Γι' αυτό το λόγο θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε ε, την ε, Βουλή την Ουγγρική καθώς και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε συνδυασμό με κοινέ συζητήσει με συζητήσει με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία υποστηρίζεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά και από τους αρχηγούς ε, κρατών ε, της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης. Ο στόχος λοιπόν είναι να δημιουργήσουμε μια αγορά στην Ευρώπη που να είναι ανοιχτή για τις επιχειρήσεις, ανοιχτή σε ό,τι αφορά τον εφοδιασμό για να δώσει τη την ε, πιο, ε, τις πιο πολλές ε, εναλλάξιμες πηγές ενέργειας και τις πιο ασφαλείς στο μέτρο του δυνατού. Πρέπει κάτι να έχουμε να προσφέρουμε πραγματικά και βέβαια ήταν μια φιλοδοξία παλαιότερη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών της και των κοινοβουλίων να οικοδομήσουν μια αγορά ενσωματωμένη, μια ευρωπαϊκή αγορά. Ε, γι' αυτό φτιάξαμε τα λεγόμενα πακέτα πρώτο, δεύτερο, τρίτο πακέτο τα οποία ως ε, στόχο είχαν να ε, εφοδιάσουν την Ευρώπη με τα απαραίτητα ούτως ώστε να έχει ένα ανταγωνιστικό επίπεδο και να δώσει στους πάντες τη δυνατότητα να υποφεληθούν από την εμπορία της ενέργειας, από την ασφάλεια της παροχής στους πάντες καθώς και την ασφάλεια των, της ζήτησης σε ό,τι αφορά αυτούς που εφοδιάζουν την Ευρώπη. Ε, επίσης η αγορά αυτή που δημιουργήσαμε είναι ολοκληρωμένη και ανοιχτή. Το θέμα όμως είναι ο εφοδιασμός των ομάδων που προέρχονται είτε προέρχονται από την Ανατολή είτε από τη Δύση ε, πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία και γι' αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό για μας στην ε, ε, Βουδαπέστη υπό την Ουγγρική Προεδρία σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δημιουργήσουμε μια καλύτερη διασύνδεση, καλύτερο δίκτυο υποδομών. Ήταν ζωτικό το θέμα αυτό για να μπορέσει να έχει βιωσιμότητα και επιτυχία είναι αυτή η αγορά. Για να έχουμε λοιπόν ένα οικονομικό σύστημα που να στηρίζεται περισσότερο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αυτό ήταν ένα πρώτο σημαντικό σημείο. Και δεύτερον, ε, τοπική κατανάλωση που να προέρχεται από τοπική παραγωγή ενέργειας. Γι' αυτό χρειαζόταν εξυγχρονισμός των παλαιότερων δομών, των υπαρχουσών δομών και ε, υπήρχαν και διάφορες επιλογές καινούργιες όπως το φυσικό αέριο και άλλες επιλογές ούτως ώστε να είναι πιο αποτελεσματική η ε, οργάνωση της αγοράς. Όλα αυτά βέβαια εξαρτώνται από την ανάπτυξη ε, του, του εφοδιασμού, του ανεξάρτητου εφοδιασμού, είτε είναι μέσα στην Ευρώπη είτε είναι εκτός Ευρώπης. Υπάρχει και το θέμα της νομοθεσίας στην Ευρώπη. Ε, δηλαδή πρέπει να δώσω σε σχέση με το θέμα αυτό της νομοθεσίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο στον τομέα της ενέργειας ένα πολύ απλό ε, μήνυμα. Πρέπει να δημιουργήσουμε ευκαιρίες. Δηλαδή να αφήσουμε τους αγωγούς και τα δίκτυα να ε, οργανωθούν κατά ένα τέτοιο τρόπο ούτως ώστε οι υπάρχοντες ανταγωνιστές να μπορούν να δουλέψουν, να ε, υπάρχουν όμως και καινούργοι οι οποίοι να μπορούν να εισαχθούν στο σύστημα και να πάρουν μέρος στο υπάρχον σύστημα. Να μην γίνεται dumping στις αγορές διότι τότε έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Να υπάρχει ανεξάρτητη διαχείριση και εξάρτητη επένδυση στο ε, δίκτυο αυτό και όλα αυτά είναι προς το συμφέρον των χρηστών. Αυτό είναι και το light motif του τρίτου πακέτου του 2009 το οποίο εφαρμόζεται την παρούσα στιγμή και εφαρμόζεται βέβαια με την συνεργασία των κρατών μελών και την ε, μεταφορά του κοινοτικού δικαίου στο εθνικό δίκαιο της ε, σχετικής οδηγίας. Είναι πάρα πολύ σκληρή δουλειά και τα αυξημένα τα καθήκοντα των ε, υπαλλήλων της Κομισιόν σε αυτό το τομέα. Ε, το εμπόριο σημαίνει ε, να εκπονηθούν κώδικες οι οποίοι να δίνουν στοιχεία για το πώς θα χρησιμοποιείται σωστά το δίκτυο, πώς θα είναι πιο εύκολη αυτή η χρήση, είτε στο Ταλίν είτε στο Πόρτο, να μπορεί κανείς να εφοδιαστεί με πετρέλαιο και αυτό σημαίνει ότι χρειάζονται ρευστότητε, χρειάζεται ευελιξία και καλύτερες τιμές στην Ευρώπη. Δεν ε, περιμένουμε βέβαια να πέσουν οι τιμές της ενέργειας στην Ευρώπη ή αλλού στον κόσμο. Το σημαντικό όμως είναι η Ευρώπη να δώσει ένα πλαίσιο στον εαυτό της, ε, ε, μια ρύθμιση ούτω ώστε να είναι δυνατόν να εισαχθούν μέσα εφοδιασμού αποτελεσματικά. Αποτελεσματικός εφοδιασμός λοιπόν με ρύθμιση και εφαρμογή αυτής της καινούργιας νομοθεσίας καθώς και ε, εκατοντάδες συστήματα διαβίβασης ε, των στοιχείων του δικτύου, ε, βελτίωση των υποδομών για να υπάρξει μια σωστή βάση για αυτόν τον ανταγωνισμό ε, και να υπάρχει ασφάλεια στον εφοδιασμό και τον ανεφοδιασμό της Ευρώπης. Όλα αυτά είναι σχέδια που αφορούν τις υποδομές. Χρειαζόμαστε υποδομές για την ανταγωνιστικότητα όλων των χωρών μας. Ε, θα πρέπει να συνδέσουμε το δυναμικό, το ενεργειακό από άκρη σε άκρη της Ευρώπης και έξω από την Ευρώπη είναι να, υπάρξει μια ποικιλομορφία στην παροχή ε, στην, στον εφοδιασμό του φυσικού αερίου να μην έχουμε ένα διάδρομο Ανατολή Δύση μόνο για τον εφοδιασμό σε φυσικό αέριο δηλαδή χρειάζεται ε, μια ποικιλομορφία. Επίσης, ε, ένας ε, άξονας βορρά-νότου για το φυσικό αέριο και για τον εφοδιασμό, ούτω ώστε να υπάρχει μια αναλλακτική λύση για τον κόσμο. Ενσωμάτωση ε, της αγοράς φυσικού αερίου που υπάρχει στην Βαλτική και πέρα από αυτό να, μπορεί να υπάρξει μια πρόσβαση για τον νότο της Ευρώπης. πρέπει να αναπτύξουμε έξυπνα συστήματα που να μπορούν να ανταποκριθούν στις νέες ανάγκες και στις νέες ρευστότητες που είναι ζωτική σημασία για την μετάδοση του φυσικού αερίου και σε επιχειρήσεις βέβαια ε, που θέλουν να, είναι, να έχουν πιο ανταγωνιστικές ε, πηγές ε, εφοδιασμού ενέργειας. Θα ήθελα κάθε κράτος μέλος να μπορεί να καταλάβει και να σχολιάσει την εθνική πολιτική, να χρησιμοποιήσει αποτελεσματικά την ενέργεια. Εάν μπορούμε να επινοήσουμε νέους τρόπους ώστε να χρησιμοποιηθεί με μεγαλύτερη ευφυΐα το όλο σύστημα από τους καταναλωτές, εάν μπορούμε να τους δώσουμε την πληροφόρηση που χρειάζονται για να χρησιμοποιήσουν το ηλεκτρικό ρεύμα και άλλες πηγές ενέργειας ε, σωστά, αυτό είναι πραγματικά θεμελιακή σημασία. Υπάρχουν πάρα πολλέ προκλήσει. Το πρώτο είναι ε, οι ρυθμίσει, σε εθνικό επίπεδο. Ε, οπωσδήποτε ο καθένας, τα εθνικά κράτη θέλουν πρώτα να εξυπηρετήσουν τα εθνικά συμφέροντά τους, αλλά υπάρχει και το ευρωπαϊκό συμφέρον. Πρέπει λοιπόν να κατανοήσουμε ότι όταν ικανοποιηθεί το, σε εθνικό επίπεδο ε, μια οργάνωση ε, ε, ευνοείται και ολόκληρη η Ευρώπη. Αυτό το είδαμε να επαληθεύεται στην κεντρική Ευρώπη και υπάρχει ανάγκη ρυθμιστών και υπάρχει ανάγκη να συμφωνήσουν ε, για τα ποσά τα οποία θα επιστρέφονται στους επενδυτές τους ώστε να μπορούν να έχουν κάποιο κέρδος ε, ε, εφόσον επενδύουν σε νέους συνδέσμους στον τομέα της ενέργειας. Σε ό,τι αφορά τη διαδικασία στην Ευρώπη έχουμε 10 με 12 χρόνια για να περάσουμε από την απόφαση ενός σχεδίου στην εφαρμογή του. Είτε πρόκειται για την παραγωγή ενέργειας, είτε για, μια νέα, για νέες γραμμές ηλεκτρικού ρεύματος, είτε για άλλες εναλλακτικέ πηγές. Τα προβλήματα λοιπόν που προκύπτουν, όπως είπε και ο πρόεδρος του ΖΕΚ, οι προκλήσεις τις οποίες αντιμετωπίζει η Ευρώπη για, την, για τον εφοδιασμό της ενέργεια είναι ζωτικό χαρακτήρα. Τόσο πολύ ε, που χρειάζεται οπωσδήποτε να βρεθούν τρόποι για να υπάρξει ασφάλεια στον εφοδιασμό, ε, για να υπάρξει ασφάλεια στην παροχή, δηλαδή κάτι οπωσδήποτε πρέπει να κάνουμε για αυτά τα ενδιάμεσα 10 με 12 χρόνια, τα οποία είναι απαραίτητα για να περάσουμε στην επόμενη φάση και για να υπάρξει εφαρμογή ε, ενός καινούριου σχεδίου. Αντί, πρέπει να δούμε τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα αυτών των νέων σχεδίων, να μεταφέρουμε όλα αυτά τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα σε τοπικό επίπεδο και περιφερειακό και να βρούμε λύσεις που να είναι αποδεκτές σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Ε, πρέπει να περάσουμε από 10 σε 12 χρόνια που είναι το, η προθεσμία σήμερα, στα 4 με 5 χρόνια πρέπει να μειώσουμε οπωσδήποτε αυτό το διάστημα. Ε, επίσης ε, υπάρχουν απαραίτητα ενεργειακά σχέδια για να διασφαλίσουν όλους τους εφοδιασμούς μας σε εθνικό επίπεδο, όλα αυτά μπορούν να αντικατοπτριστούν στο σχέδιο το γενικότερο που αφορά ε, το φυσικό αέριο και τον ηλεκτρισμό ε, θα χρηματοδοτηθούν αυτά τα σχέδια μερικά άλλα όμως δεν θα χρηματοδοτηθούν και ε, πρέπει να υπάρξει μια προσπάθεια να δοθούν χρηματοδοτήσεις αντίστοιχες ιδιωτικές που να αντιστοιχούν στις επενδυτικές ανάγκες. Ε, ίσως ε, όταν δεν μπορεί ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός να ανταπεξέλθει να πρέπει ο εθνικός προϋπολογισμός να μπορεί. Τώρα ε, υπάρχει επίσης και ένα ουσιαστικότατο σημείο δηλαδή για να γίνει ε, ε εφοδιασμός για να γίνουν τα ευφυή δίκτυα ε, θα πρέπει να μπορέσουμε να διαχειριστούμε τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούν τον ίδιο ηλεκτρισμό στις κατοικίες, στα σπίτια με έναν τρόπο με τον οποίο να ωφελούνται για να μπορούμε να προβλέψουμε και τις ε, δυνατότητες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη σαν σύνολο. Αυτό απαιτεί επενδύσεις πάρα πολύ ακριβές για τα επόμενα 40 με 50 ή ακόμα και 60 χρόνια. Θα ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την υποστήριξη υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, να καταρτιστεί ένας οδικός χάρτης ε, για τα επόμενα χρόνια ε, και θα το παρουσιάσουμε αυτό το σχέδιο το Νοέμβριο του φετινού έτους. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. darf mich bedanken ganz herzlich für diesen Einstieg und Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσίαση, την εισαγωγή παρουσίαση που κάνατε. Στρέφομαι προς το Συμβούλιο για να ακούσουμε κάποιον εκπρόσωπο τη της Ουγγρικής ε, Προεδρίας και συγκεκριμένα ο κ. Πάλκοβας, ο Υπουργός Ενέργειας κυβέρνηση. θα πάρει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε Μπούζε και Γενική Διευθύντα. Το μικρόφωνο σας. Yes. Can you hear me, please? Yeah, okay.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 ε, Αξιότιμε Πρόεδρε Μπούζεκ, κύριε Γενική Διευθυντά, κύριε Ευρωβουλευτές, κυρίε και κύριοι, είναι μεγάλη χαρά για μένα που βρίσκομαι εδώ και που εκπροσωπώ την Ουγγρική Προεδρία. Τα θέματα έχουν που έχουν τοποθετηθεί στην ημερήσια διάταξη έχουν σχέση με τα... ε, τις δραστηριότητες της Προεδρίας μας σε σχέση και με τις υποδομές. Θα ήθελα να κάνω μερικές παρατηρήσεις και να σας πω τι έχει γίνει και τι απομένει να γίνει στους επόμενους, στις επόμενες εβδομάδες της Προεδρίας μας. Όπως ήδη τονίστηκε από πολλούς, η ενέργεια είναι από τα πιο περίπλοκα θέματα, τις μεγαλύτερες προκλήσεις σήμερα για να εξασφαλίσουμε ε, την ε, ευημερία, την εθνική ασφάλεια πρέπει να βελτιώσουμε ε, την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού και την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης ενώ βεβαίως θα διατηρήσουμε ένα φόρο βιώσιμο περιβάλλον. Αυτό το θέμα έχει μεγάλη προτεραιότητα για την Προεδρία μας. Είχαμε δράσεις για την διατηρησιμότητα, την ασφάλεια ε, και τις ολοκληρωμένες εντεταγμένες αγορές Πρόκειτο για δύσκολο έργο και ε, συμβάλαμε όμως νομίζω στους στόχους σχετικά με την ε, διαφορία και την ε, διατηρησιμότητα. Θέλαμε στρατηγικές μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες. Ο στόχος αυτός ενθαρρύνθηκε από το πρώτο Συμβούλιο της 4ης Φεβρουαρίου όπου τα μέλη διακήρυξαν τη δέσμευσή τους για ένα μια πραγματικά ενιαία αγορά ε, ηλεκτρισμού και αερίου μέχρι το 2014, εκτός ώστε κανένα κράτος να μην είναι απομονωμένο από αυτήν την αγορά ε, από το 2015. Πρέπει να τονιστεί περισσότερο η ενεργειακή αποδοτικότητα ε, και οι εξωτερικές σχέσεις ούτως ώστε να επιτύχουμε τους στόχους του 2020. Με τις κατευθυντήριες γραμμές του Συμβουλίου υιοθετήθηκαν συμπεράσματα για την ανακοίνωση ενέργειας 2020 ε, για τον τομέα της ενέργειας και επιτύχαμε στις 24 Φεβρουαρίου στο Συμβούλιο Ενέργειας να ενισχύσουμε και να επανεπιβεβαιώσουμε τα αποτελέσματα και τους στόχους του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Σχετικά με την πρακροπρόθεσμη στρατηγική Ουγγρική Προεδρία θέλει να αρχίσουμε ε, συζητήσεις για τον οδικό χάρτη 2020 με το Συμβούλιο Γκέρνινγκ στην Ουγγαρία στις αρχές αυτού του μήνα. Πιστεύουμε ότι οι συζητήσεις έδωσαν μεγάλη όθηση στην οριστικοποίηση των προτάσεων της Επιτροπής. Σε σχέση με την αηφορία, την διατηρησιμότητα, είχαμε τον φάκελο με τον πρόγραμμα για την ενεργειακή απόδοση. Μετά από μια ενδελεχή συζήτηση στην ομάδα εργασίας στις 10 Ιουνίου ε, θα υιοθετηθούν συμπεράσματα στο Ενεργειακό Συμβούλιο σχετικά με την ασφάλεια και την επάρκεια του εφοδιασμού. Συζητήσαμε την ανακοίνωση για τις διεθνείς σχέσεις στον τομέα της ενεργειακής πολιτικής όπως και την κατάσταση προόδου ε, σχετικά με την παραγωγή αερίου υπεράκτια ασχοληθήκαμε με την εξωτερική ε, διάσταση, ε, την ενεργειακή συζήτηση. Ήταν μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων σχετικά με το θέμα αυτό, σχετικά με τον στόχο της ενιαίας ολοκληρωμένης αγοράς. Ε, ένας από τους στόχους μας ήταν να έχουμε μια συμφωνία για την ρύθμιση, για την ε, μεταφορά, την θαλάσσια μεταφορά ενέργειας. Στην ε, Συμβούλιο του Ιουνίου μπορεί να καταλήξουμε σε πολιτική συμφωνία ε, μετά από συζητήσεις στην ομάδα εργασίας και εν ώψη του τριμερούς διαλόγου ανάμεσα στην Επιτροπή, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο θα έχουμε ελεύθερες τριμερείς συζητήσεις στις 16, 23, 29 Ιουνίου ούτως ώστε να έχουμε πολιτική συμφωνία. Η τελική προσαρμογή του κανονισμού από το Κοινοβούλιο αναμένεται το Σεπτέμβριο. Τα συστήματα υποδομών της Ευρωπαϊκής Ένωση ίσως να ήταν ε, το πιο σημαντικό θέμα στην ημερήσια μας διάταξη. Δεν μας εκπλήσει αυτό. Η νέα ενεργειακή στρατηγική από το 2011 στο το 2020, όπως και η Σύνοδος Κορυφής Ενεργειακή του Φεβρουαρίου, απέδωσαν ιδιαίτερη προσοχή στην ανάπτυξη των υποδομών, ούτως να υπάρξει ένα μοντέλο για αυτήν την δεκαετία για υποδομές ε, και η κατάργηση της απομόνωσης οποιαδήποτε κράτους από τις αγορές. Η Επιτροπή, η οι ε, Υπουργοί Ενέργειας υιοθέτησαν ανακοίνωση τον Φεβρουάριο σε σχέση με τις προτεραιότητες και την χρήση των πιο αμέσων παραδειγμάτων. Έχουμε μια υψηλού επίπεδου ομάδα εργασία για τις χώρες Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης για να προσδιοριστούν οι ανάγκες και προτεραιότητες σε υποδομέ της περιοχή και να υπάρξει ε, μια διασύνδεση αποτελεσματική βορρά-νότου. Η Προεδρία μας επίση. Ε, οργάνωσε σε συνεργασία με την Επιτροπή μια διάσκεψη επιλού επίπεδου για τις ενεργειακές ευρωπαϊκές υποδομές ε, πριν από μία εβδομάδα οι κυβερνήσεις, οι ρυθμιστές, οι φορείς μεταφοράς, οι οικονομικοί οργανισμοί και άλλοι εμπλεκόμενοι συζήτησαν τις βασικές προκλήσεις και δυνητικές λύσεις για τα προβλήματα σχετικά με την κατασκευή ενεργειακών υποδομών. Με τις παρουσιάσεις είδαμε ποιες είναι οι εξελίξεις, οι τεχνολογικές που επιτρέπουν ε, μηχανισμούς για την μεταφορά ε, και την κατανομή του κόστους. Θα ήθελα και πάλι να σας ευχαριστήσω που βρίσκεστε εδώ σε αυτήν την μεικτή συνεδρίαση Επιτροπών Εθνικών Κοινοβουλίων και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την βελτίωση του ενεργειακού εφοδιασμού. Ε, περιμένω με ενδιαφέρον ε, τα συμπεράσματα σχετικά με τις διαδρομές ε, διότι νομίζουμε ότι ο τομέας της ενέργειας και η ανάπτυξη των υποδομών είναι μια γέφυρα που θα επιτρέψει στην Ευρώπη να γίνει πιο ανταγωνιστική, πιο ασφαλής και να έχει ένα μέλλον πιο καθαρό. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Äh, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσοι συμμετέχουν στη σημερινή μεικτή συνεδρίαση και να ευχαριστήσω όλους ιδιαίτερο την ε, Ουγγρική Προεδρία που ανέλαβε την πρωτοβουλία. Ευχαριστώ επίσης και το Ουγγρικό Κοινοβούλιο για την πρωτοβουλία διοργάνωση αυτής της ε, μικτής ε, συνεδρίας σας. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους από τα Εθνικά Κοινοβούλια και ευχαριστώ και τους εκπροσώπους της ε, Ουγγρικής ε, Προεδρίας που διότι έχει ως στόχο τον ε, ενεργειακό εφοδιασμό σε προσιτές τιμές όντως ήταν ένας από τους βασικούς στόχους της Προεδρίας σας. Θεωρώ ότι είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι θα ακολουθήσει την ίδια ρότα και η επερχόμενη Προεδρία, η Πολωνική Προεδρία. Ε, πάντως ε, για μας ε, δεν αλλάζει τίποτα στο ρόλο του νομοθέτη. Ο στόχος μας εξακολουθεί να είναι να κατοχυρώνουμε την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού, να έχουμε καλύτερη απόδοση στη χρήση της ενέργειας, να αναπτύξουμε νέες τεχνολογίες, ε, να χρησιμοποιούμε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, να υπάρχει καλύτερη διασυνδεσιμότητα των δικτύων, γιατί αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για την εσωτερική αγορά. Αυτό θα είναι εξάλλου και μία από τις βασικότερες προκλήσεις και ο Πρόεδρος το ανέφερε, πρέπει να καλύψουμε τι ενεργειακέ μας ανάγκε, όχι μόνο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο, διότι έχουν όλη την τάση να πιστεύουν ότι θα χρειαζόμαστε, λένε, και περισσότερη ενέργεια, Θα χρειαστούν λοιπόν εθνικές αποφάσεις, ώστε να προσανατολιστούμε προς ε, μορφές ενέργειας που θα εξυπηρετήσουν τις ανάγκες μας. Χρειάζεται έρευνα, λοιπόν, έρευνα ακόμη και στον τομέα της ε, ε, σχάσης. Πώς μπορούμε λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο να έχουμε ένα εύρυθμο σύστημα, οι τιμέ να είναι προσιτές ακόμη και για τα μεσαία εισοδήματα, αλλά ακόμη και για τα χαμηλά εισοδήματα να εξασφαλίσουμε ενεργειακό εφοδιασμό. Πώς μπορούμε επίσης να επιτύχουμε τιμέ αποδεκτές από την βιομηχανία. Πολλά κεντρικά ζητήματα πρέπει να εξετάσουμε και βασική πρόκληση για μας ε, θα είναι να συνδυάσουμε τους πολιτικούς στόχους ε, με τους ε, νομοπαρασκευαστικούς μας στόχους και να ρυθμίσουμε οποιαδήποτε προβλήματα ανακύψουν. Με ποιο τρόπο μπορούμε να μεταφέρουμε την αιωλική ενέργεια στα κέντρα κατανάλωσης. Ε, Φερρυπίν, πώς μπορούμε να αναπτύξουμε φιέστερα δίκτυα, πώς ε, να δημιουργήσουμε κέντρα αποθήκευσης της ενέργειας. Ε, με ποιο τρόπο μπορούμε να αποφύγουμε τη ρήξη τις ε, διαμάχες ανάμεσα στους, πολιτικ... Ε, στους πολιτικούς στόχους και τους νομοθετικούς στόχους. Μια άλλη μεγάλη πρόκληση είναι να βρούμε επαρκείς πόρους και για την έρευνα αλλά και για την δημιουργία νέων ε, ρηξικέλευθων τρόπων για την κατοχήρωση της, ε, του ενεργειακού μας ε, εφοδιασμού. Χρειάζονται λοιπόν μακρόπνοες αποφάσεις πέρα από τον άμεσο σχεδιασμό, μια σταδιακή προσέγγιση που θα περνάει σίγουρα από τη δημιουργία ε, συστημάτων, εφιών συστημάτων ενέργειας για να είναι διαθέσιμη η ενέργεια που χρειαζόμαστε Χρειαζόμαστε ευφιέστερη υποδομή για να ε, ε, επιτύχουμε καλύτερη ισορροπία ανάμεσα στην προσφορά και στη ζήτηση. Ε, είναι επίσης σημαντικό να δούμε κατά πόσο θα αυξήσουμε το ποσοστό των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μέσα στο ενεργειακό μείγμα της Ένωσης, χωρίς όμως να υπονομεύσουμε ούτε την ανταγωνιστικότητά μας, ούτε την ασφάλεια ε, του ενεργειακού ε, εφοδιασμού. Αυτό θα καταστεί δυνατό μόνο αν διευρύνουμε τα δικτύα μας, τα συνδέσουμε με καλύτερο τρόπο και τα καταστήσουμε ευφιέστερα. Χάρη στη συνθήκη της Λισαβόνας μπορούν τώρα να διαδραματίσουν σημαντικότατο ρόλο και τα Ευρωπαϊκά Κοινοβούλια για όλους τους τομείς όπου ε, νομοθετεί και παρεμβαίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο ενδιάμεσο διάστημα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βρίσκεται πλέον στο κέντρο, στην καρδιά της νομοπαρασκευαστικής διαδικασίας σε βάση του άρθρου Τη της νέας συνθήκης, συγκεκριμένα τα ενεργειακά ζητήματα, ε, ανήκουν πλέον στο πεδίο που έχει ενισχυμένε νομοθετικέ αρμοδιότητε στο Κοινοβούλιο. Είμαστε σύνομοθετες πλέον για το ζήτημα αυτό. και ε, αυτά τα επόμενα χρόνια να αντιμετωπίσουμε βασικές προκλήσεις και γι' αυτό θα χρειαστεί μια στενή συνεργασία ανάμεσα στο Κοινοβούλιο, τα κράτη-μέλη, τις ε, τοπικές αυτοδιοικητικές αρχές και φυσικά με τους συναδέλφους μας από τα Εθνικά Κοινοβούλια. Ε, αναμφισβήτητα, το θέμα της επικουρικότητας θα πρέπει να θεωρηθεί εξίσου σημαντικό όπως και η σημασία της κοινή προσέγγισης αν δεν θέλουμε να απομακρυνθούν οι εκλογές μας από εμά. Θα ήθελα τώρα να σας ε, μιλήσω εντάχει για αυτά που έχουν γίνει στην Επιτροπή Ήτρα. Τα 45 μέλη της Επιτροπής Βιομηχανίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, έχουν καταβάλει ήδη σημαντικότητα τις προσπάθειες ε, για να ενισχύσουν την αποτελεσματικότητα της ενίας αγοράς, να προαγάγουν την εξοικονόμηση και την αποδοτικότερη χρήση της ενέργειας, την δημιουργία ευφιέστερων δικτύων και την εξέβρεση νέων ενεργειακών πηγών. Όλες αυτές οι παράμετροι είναι απαραίτητες για να δημιουργήσουν ε, μία ενιαία αγορά ενέργεια και τον τελευταίο χρόνο διαδραματίσαμε σημαντικό ρόλο για την υιοθέτηση νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια του εφοδιασμού σε φυσικό αέριο. Εδώ στο Κοινοβούλιο έγινε επίση σημαντικότατη συζήτηση ε, για τι ε, επιδοτήσει ε, τη Ένωση για την έρευνα για νέε πηγέ ενέργεια και επίση σχετικά με την ολοκλήρωση τη ενεργειακή αγορά και την διαφάνεια των αγορών. Έχουμε ήδη καταθέσει πρόταση είναι ένα θέμα πάρα πολύ σημαντικό για τους καταναλωτές. Η Επιτροπή βιομηχανία του Κοινοβουλίου αλλά και συνολικότερα το Κοινοβουλίο τόνισαν πόσο σημαντικό είναι να έχουμε ταχύτατη πρόοδο αν θέλουμε να ε, υλοποιήσουμε τους στόχους που είχαμε θέσει μέχρι το 2020, δηλαδή να έχουμε ε, αποδοτικότερη ε, χρήση της ενέργειας μέχρι το 2050 στα πλαίσια του Γενικότερου Στρατηγικού Σχεδιασμού. Επίσης, μιλήσαμε Συζητήσαμε για την ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι το 2020. Θα μας επιτρέψει να έχουμε μια μακρόπνοη θεώρηση για την περίοδο που θα καλύπτει μέχρι και το 2050 αυτή η προσέγγιση συνεπάγεται ότι θα έχουμε και ε, βρέχει μέσω πρόθεσμους ε, ενεργειακούς στόχους ε, και μικρότερα προγράμματα. Η, ενεργεια, η αποδοτική χρήση πάντως της ενέργειας είναι ένα από τα βασικά προβλήματα που μας απασχολούν. Έχουμε συνεργαστεί στενά με τον Επίτροπο Έτιγκερ. Σε σχετικές εκθέσει έχουμε απαριθμίσει όλε τι προτεραιότητε του Κοινοβουλίου και τον Ιούλιο θα εγκριθεί αυτή η έκθεση του Κοινοβουλίου ε, για το θέμα αυτό. Επίσης, ε, θα πρέπει να διευκολύνουμε τις επενδύσεις. Ο εξυγχρονισμό είναι επίσης ένα άλλο σημαντικότατο βήμα εξυγχρονισμό δηλαδή των υποδομών και των ε, δικτύων. Η Επιτροπή λοιπόν βιομηχανία επιθυμεί να ε, συμβάλλει ενεργά ε, στην υλοποίηση ε, της ενεργειακής στρατηγικής της Ένωσης. Κατά πάσα πιθανότητα θα καταθέσει πρώτα τον Οκτώβριο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για αυτό το θέμα. Βλέπετε λοιπόν πόσο ευρύ είναι το φάσμα των κατοικών που έχει η Επιτροπή μας. Ούτως ή άλλως αυξανόμενη σημασία του ζητήματος. Τα τελευταία χρόνια λοιπόν έχει αυξηθεί και ο φόρτος εργασίας μας. Ε, προφανώς ε, θα πρέπει να είμαστε φιλόδοξοι, αλλά όπως όλοι γνωρίζουν, ε, ταυτόχρονα θα πρέπει να είμαστε και ρεαλιστές. Όχι μόνο φιλόδοξοι, θα πρέπει να σεβαστούμε αυτό το παραδοσιακό τρίγωνο, δηλαδή αηφορία, ασφάλεια και εύλογες τιμές. Χαίρομαι ιδιαίτερος λοιπόν που οργανώσαμε την σημερινή μεικτή συνεδρίαση ούτω ώστε να μην συνεργαζόμαστε μόνο με την Επιτροπή και το Συμβούλιο, αλλά και με τι εθνικέ κυβερνήσει και πάνω απ' όλα με του συναδέλφου μα από τα εθνικά κοινοβούλια. Μετά από αυτές τις σύντομες εισαγωγικέ παρατηρήσεις ε, θα δώσω και πάλι το λόγο στον ε, συνάδελφο Ρογκάν που ήδη ανακοίνωσε θα ήθελε να μας δώσει κάποια συγκεκριμένα παραδείγματα από την αντίστοιχη Επιτροπή του Ουγγρικού Κοινοβουλίου. Κυρίες και κύριοι Ευρωβουλευτές, κυρίες και κύριοι βουλευτές των Εθνικών Κοινοβουλίων, το θέμα της σημερινής συζήτησης αναφέρεται σε ενεργειακούς διαδρόμους και ως εισαγωγή θα ήθελα να πω ότι εδώ και μερικά χρόνια διαπιστώσαμε τη σημασία τους όταν τη στιγμή όπου το ρωσικό αέριο υπέφερε όπου ο εφοδιασμός από ρωσικό αέριο υπέφερε. Είδαμε τη σημασία τους για την ενεργειακό εφοδιασμό και την σημασία της αγοράς ενέργειας. Τότε το Συμβούλιο του Φεβρουαρίου της Ουγγρικής Προεδρίας προσπάθησε ούτως ώστε το 2015 αυτή η κατάσταση να μην επαναληφθεί. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε τη διασύνδεση ανάμεσα στους διάφορους ενεργειακούς διαδρόμους. Πρόκειται για ένα θέμα που συζητείται σε διάφορα φόρα και εκτός από το διάδρομο του Νότου υπάρχουν και οι διάδρομοι του Βορρά που συνδέουν τη Βαλτική με τη Βόρεια Θάλασσα οι διάδρομοι οι οποίοι συνδέουν τους καταναλωτές ε, του Νότου με το Βορρά και αυτούς του Βορρά. Αυτό αντιπροσωπεύει τεράστιες επενδύσεις. Πρέπει λοιπόν να προβλέψουμε σημαντική χρηματοδότηση. Εφόσον πρόκειται για τη χρηματοδότηση, υπάρχει ένα θέμα το οποίο τίθεται βεβαίως. Θα υπάρχει μια κοινοτική χρηματοδότηση. Πρόκειται για τη δημιουργία, τη διαμόρφωση μιας ευρωπαϊκής αγοράς, αλλά εφόσον πρόκειται για χρηματοδότηση ευρωπαϊκή, αυτό θα γίνει παρά μόνο κατόπιν ενδελεχούς και προσεκτικής μελέτης του θέματος και όλου του, των επιπτώσεων του πάντως. Η χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα είναι απαραίτητη για να υπάρξει αυτή η διασύνδεση ως προς τις επιλογές των ε, επενδύσεων και αυτή η συζήτηση θα είναι πάρα πολύ σημαντική. Το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή έχουν πάρα πολλές ιδέες να ανταλλάξουν και μετά θα πρέπει να γίνουν στρατηγικές επιλογές που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν πραγματικές διασυνδέσεις στην Ευρώπη βραχυπρόθεσμα. Σε 10 ή 15 χρόνια δεν θα έχουμε τον απαιτούμενο χρόνο για να έχουμε όλες τις διασυνδέσεις που χρειάζονται για τον εφοδιασμό ε, της ευρωπαϊκής αγοράς. Λόγω του ύψους των προβλεπωμένων επενδύσεων χρειάζεται χρηματοδότηση της Ένωσης αλλά και χρηματοδότηση που θα προέλθει από την αγορά. Θα προέρχεται από την αγορά. Και εδώ και πάλι το ίδιο θέμα τίθεται. Ποιος θα πληρώσει το τίμημα και για τους καταναλωτές. Το έργο των ρυθμιστών είναι ιδιαίτερα σημαντικό και το έργο αυτό ανήκει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή που θα πρέπει να προσδιορίσει ένα γενικό πλαίσιο ε, κατανομής του κόστους. Ένα γενικό πλαίσιο το οποίο θα μας επιτρέψει να δούμε ποιες είναι οι επενδύσεις που είναι δικαιολογημένες. Κάθε επένδυση θα μπορούσε να επιβαρύνει τους καταναλωτές αν τους εξηγήσουμε καλύτερα ότι θα μειωθεί η ενεργειακή εξάρτηση, ότι θα υπάρχει μια αποδοτική ενεργειακή πολιτική ούτω ώστε η ενέργεια να είναι λιγότερο ακριβή. Θα δοθούν εγγυήσεις στους καταναλωτές και ο ρόλος του ρυθμιστή είναι ακόμη πιο σημαντικός διότι θα πρέπει να λάβει υπόψη όλα αυτά τα στοιχεία και να βρει μια ισορροπία ανάμεσα στα συμφέροντα των καταναλωτών, των προμηθευτών και ούτω καθεξής. Βεβαίως, ξέρω πολύ καλά ότι αυτή η κατανομή του κόστους ανάμεσα στην αγορά, τους χρήστες, την Ευρωπαϊκή Ένωση θα προκαλέσει μεγάλη συζήτηση, αλλά το ύψος των ε, αναγκαίων επενδύσεων απαιτεί την ύπαρξη ενός ρυθμιστή. Θα το δούμε στα επόμενα χρόνια. Εξάλλου, σε σχέση με το θέμα αυτό, λέμε ότι για να ρυθμιστούν οι ευρωπαϊκές αγορές θα πρέπει να βρεθούν επενδύσεις μακροπρόθεσμες με ένα μηχανισμό παρακολούθησης, εποπτείας για να ε, δημιουργηθεί αυτός ο μηχανισμός χρειάζεται χρόνος για να επανέλθω στο θέμα μου θα πρέπει να λάβουμε υπόψη αυτό το σημείο εκκίνησης που είναι βασική προϋπόθεση. Θα μιλήσουμε σε λίγο για τις, ε, τους ενεργειακούς διαδρόμους. Δεν ε, θα αναφερθώ σε αυτούς τώρα για να μην αναμίξουμε τα διάφορα σημεία της ημερήσιας διάταξης εφόσον ε, θα έχουμε την ευκαιρία να επανέλθουμε στο θέμα αυτό. Αυτές είναι οι ιδέες που ήθελα να υποβάλω για την ώρα. Ευχαριστώ πολύ. Ε, θα ήθελα τώρα τελειώσαμε με το εισαγωγικό μέρος και θα αρχίσουμε με το θέμα αυτό καθεαυτό ε, θα σας παρακαλούσα να ξανααναλάβετε την Προεδρία. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να επισύρω την προσοχή των συμμετεχόντων πάνω σε ορισμένα σημεία. Το πρώτο θέμα είναι συνεπώς η ενεργειακή διάδρομη. Δύο πράγματα είναι σημαντικά για τους ευρωβουλευτές και τους εθνικούς βουλευτές. Θα έχει τρία λεπτά ο κάθε παρεμβαίνων για κάθε παρέμβαση. Μετά θα προσπαθήσουμε να έχουμε έναν κατάλογο μεικτών ε, παρεμβενόντων. Θα έχουμε δύο από τα εθνικά κοινοβούλια, έναν από το Ευρωκοινοβούλιο και θα έχουμε την διαδικασία της μπλε κάρτας που μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Νομίζω ότι οι περισσότεροι από εσά γνωρίζετε αυτή τη διαδικασία. Αν θέλετε να την χρησιμοποιήσετε θα κάνω ό,τι μπορώ για να συντονίσω καλά αυτή τη διαδικασία με τις μπλε κάρτες. Είχαμε προβλέψει στις 16 και 15 μια διακοπή για καφέ 15 λεπτών. Εφόσον έχουμε καθυστέρηση σας προτείνω να μην κάνουμε τη διακοπή. Με τον τρόπο αυτό θα μπορέσουμε να έχουμε την πρώτη μας συζήτηση μέχρι τις 16 και 30. Το πρώτο άτομο στον κατάλογο των ομιλητών είναι ο κύριος ε, Καζολή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 την ε, Ιταλική Γερουσία και θεωρώ ότι είναι θεμελιακό να εξακολουθήσουμε τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως για να αυξήσουμε την ασφάλεια του εφοδιασμού ε, πέρα από τα σύνορα. Η χώρα μου η Ιταλία πάντα προσπάθησε να έχει και διπλωματικούς δεσμούς και φυσικούς ούτως ώστε να μπορεί να έχει μια καλύτερη επικοινομορφία στον εφοδιασμό. Ενέργεια Το ευρωπαϊκό σύστημα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι ανέκαθεν υπήρξε το πιο αποτελεσματικό και θα ήθελα ακόμα να πω περατώντας την παρέμβασή μου ότι πρέπει να είμαστε πάρα πολύ ε, προσεκτικοί στην συμφόρηση που μπορεί να παρουσιάζουν τα εθνικά δίκτυα. Μπορεί να υπάρχουν εξαιρετικοί διάδρομοι ε, μεταξύ κρατών μελών αλλά να μην υπάρχουν σε εθνικό επίπεδο. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να λάβω το λόγο εξ ονόματος της Οικονομικής Επιτροπής της Γαλλικής Βουλής. Είμαστε υπέρ της διασύνδεσης των δικτύων πρέπει να σας πω, διότι έτσι θα βελτιστοποιήσουμε τους πόρους μας, αλλά και θα κατοχυρώσουμε την ασφάλεια του εφοδιασμού. Ε, πέρα από αυτό πιστεύουμε ότι πρέπει να επαληθεύσουμε την συμβολή της κάθε χώρας και την προσπάθεια που καταβάλει για να σεβαστεί τις συμφωνίες που γίνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη διατήρηση του περιβάλλοντος και την προστασία του περιβάλλοντος μας. Πρέπει να υπάρξουν πολλαπλές πηγές εφοδιασμού για να μην είμαστε εξαρτημένοι σε επίπεδο εφοδιασμού και να έχουμε ε, πλούσια δίκτυα. Επίσης ε, πιστεύουμε ότι χρειάζεται αλληλεγγύη μεταξύ των διαφόρων χωρών της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τα εφή δίκτυα τώρα είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο για τις ανανεώσιμες ενέργειες ε, οι οποίες χρησιμοποιούνται εναλλακτικά και πρέπει ε, ελπίζω να έχουμε μια καλύτερη κατοχήρωση της ασφάλειάς τους. Πέρα από αυτό κύριε Πρόεδρε θα ήθελα να μιλήσω για την πρόθεση της έρευνας. Η προαγωγή της έρευνας είναι απαραίτητη αν θέλουμε να εστιάσουμε τις προσπάθειές με, τις, με μια αμοιβαία στρατηγική αντιμετώπιση ούτως ώστε η Ευρώπη να μπορέσει να ικανοποιήσει τη μεγαλύτερη δυνατή φιλοδοξία της. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Είχα κάνει λάθος στην σειρά ε, ο κύριος Ανδράς Λαπισκή είχε ζητήσει το λόγο πρώτος νομίζω. Ο κύριος λοιπόν Ανδράς Αρατσκή ε, εφόσον ξεκίνησε η συζήτηση θα λάβει το λόγο αργότερα και ζητώ συγγνώμη πραγματικά Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Γενική Διευθυντά. Υπάρχουν πάρα πολύ σημαντικά θέματα τα οποία αναφέρθηκαν. Ε, κύριε Πρόεδρε, δεν θέλω να τα επαναλάβω και να καθυστερήσω την ε, σημερινή συζήτηση. Θα ήθελα να πω ότι Υπάρχει το εξής στοιχείο τον Μάρτιο του 2007 ενέκρινε το Ευρωπαϊκό ε, Κοινοβούλιο ένα κείμενο για την ε, ασφάλεια του εφοδιασμού σε ενέργεια που είναι πάρα πολύ σημαντικό για τη συζήτηση που διεξάγεται σήμερα. Μιλού, αυτό το κείμενο θεσπίζει ε, τα καθέκαστα σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο για να μπορούμε μια μέρα να έχουμε μια σωστή εφαρμογή του. Το 2010 οργανώθηκε μια Επιτροπή η οποία ενέκρινε αυτές τις θέσεις. Γίνεται λόγος για τις υποδομές ενέργειας, για το σχεδιασμό, για τη διαχείρισή τους και υπάρχει ένα ψήφισμα το οποίο ζητά να υπάρξει ποιοτική αλλαγή στην περισυλλογή επ' αυτών των θεμάτων. Για να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια θετική αλλαγή πιστεύουμε ότι χρειάζεται το θέμα της ε, ασφάλειας εφοδιασμού και ανεφοδιασμού να είναι κάτι το δεδομένο, σε, κάτι το κεκτημένο σε εθνικό επίπεδο γιατί αυτό είναι ένα πραγματικό εθνικό πρόβλημα είναι ένα πραγματικό κοινωνικό αν θέλετε πρόβλημα στην ε, Ουγγαρία είχαμε την αρνητική εμπειρία είχαμε δει ποιες είναι οι μεγάλες επιπτώσεις της, ε, της έλλειψης εφοδιασμού. Τι αντίκτυπος υπάρχει στον πληθυσμό που υπέφερε ακριβώς τις συνέπειες γιατί δεν είχαμε σκεφτεί σωστά ή δεν είχαμε σκεφτεί αρκετά τα θέματα της κατοχήρωσης της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού. Και τελικά ολόκληρη η κοινωνία πρέπει να πούμε ε, ε, υπέστη αυτά τα δεινά, πλήττεται εάν υπάρξει πρόβλημα εφοδιασμού ενέργειας. Πρέπει λοιπόν τα κράτη-μέλη να ξέρουμε ότι έχουν τη, δική τους ασφάλεια εφοδιασμού και μετά από τα εθνικά κράτη πρέπει να ασχοληθούμε με την ασφάλεια ολόκληρης της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Το πρόβλημα αυτό δεν γνωρίζει σύνορα. Βέβαια, μια κοινή ενεργειακή αγορά είναι μια απαραίτητη προϋπόθεση πραγματικά απαραίτητη για να μπορούμε να συνεχίσουμε. Θα συνεχίσουμε λοιπόν την ανάπτυξη των εθνικών δικτύων και θα δημιουργήσουμε αυτούς τους ενεργειακούς ε, ε, διαδρόμους με ε, διασυνοριακές διασυνδέσεις ενσωματώνοντας και συνέχεια νέους καινούριου ενεργειακούς διαδρόμους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να λάβουμε υπόψη μας τα στοιχεία αυτά. Θέλουμε ευφυή δίκτυα τα οποία πρέπει να είναι πιο αποτελεσματικά, να επιτρέπουν την εξοικονόμηση ενέργειας και να είναι σε θέση να προσαρμοστούν στις ανανεώσιμες ενέργειες ούτω ώστε να μπορέσει να υπάρξει αποθήκευση της ενέργειας και ε, διανομή εκ των υστέρων στους καταναλωτές. Το φετινό είδαμε ότι τα σχέδια είναι πολλά Έχουμε σχέδια, έχουμε ιδέες, καλές ιδέες, καινούργιε ιδέες, αλλά όπως είπε και ο Πρόεδρος, μας χρειάζεται μια συνολική πολιτική, μας χρειάζεται ένα σύστημα ολοκληρωμένο και μέσα στα πλαίσια αυτού του συστήματος πρέπει να επιλέξουμε τα καταλληλότερα σχέδια, τα επαρκέστερα, τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να κατανοήσουν ότι η ασφάλεια του εφοδιασμού και η ενεργειακή διάδρομη δεν είναι ένα θέμα ανταγωνισμού μεταξύ των κρατών μελών της Ευρώπης. Είναι το θέμα του δικού μας ευρωπαϊκού και κοινού συμφέροντος το διακύβευμα. Γι' αυτό πιστεύουμε ότι πρέπει να έχουμε ένα κοινό όραμα επί της ε, ουσίας και πρέπει να ξέρουμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντική η απόφαση του Συμβουλίου του Φεβρουαρίου που μας δίδει τέσσερα χρόνια για να δημιουργήσουμε μια πραγματική αγορά φυσικού αερίου, πετρελαίου και ηλεκτρικού ρεύματος ε, στην Ευρώπη ούτω ώστε να μπορέσουμε μέσω πρόθεσμα να ε, γίνουμε ανεξάρτητοι, να σταματήσει πλέον αυτή η εξάρτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα εφοδιασμού ενεργειακού. Αυτές οι ενεργειακές νησίδες οι οποίες υπάρχουν και συνεχίζουν να υπάρχουν μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να καταργηθούν. Επίσης πρέπει να πάψουν να υπάρχουν αυτά τα ενεργειακά διέξοδα, αυτές οι αδυναμίες προσαρμογής στους ενεργειακούς διαδρόμους. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα διότι πρέπει να τους συντηρήσουμε, πρέπει να μπορούμε να τους συντηρήσουμε και να, να υπάρχει διαρκή συντήρηση ε, γι' αυτό ε, μέσα στα διέξοδα που αντιμετωπίζουμε πρέπει να κατανοήσουμε ότι φτάνουμε σε πολύ δύσκολες καταστάσεις αυτό όπως η κατάσταση της Ουγγαρίας ε, τον χειμώνα του 2009. Για να κατοχυρώσουμε λοιπόν την ασφάλεια εφοδιασμού ενέργειας προβλέψαμε την δημιουργία δικτύων από το βορρά στο νότο με συνδέσεις από το, στην κεντρική Ευρώπη από το βορρά ως στο Νότο και έχουν ήδη ληφθεί μέτρα, έχει ληφθεί μια σειρά μέτρων στη χώρα μας για διασυνδέσεις για παράδειγμα στα σύνορα με τη Ρουμανία ε, και με την Κροατία άλλο ένα παράδειγμα είναι έτοιμες αυτές οι εγκαταστάσεις από το πέρας του 2010 και έχουν γίνει μεγάλα έργα τα οποία ε, συνεχίζονται δεν έχουν ακόμα περατωθεί ούτω ώστε να ανοίχτεί μια άλλη γραμμή πέρα από την γραμμή βορρανότου. Εμείς ε, έχουμε υπογράψει τα συμβόλαια και προχωρούμε. Αυτό θέτει και μια σειρά ε, προβλημάτων, ερωτημάτων μάλλον μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα σας δώσω μερικά παραδείγματα η σύνδεση του Sunstream με τον Αμπούκο. Είναι δίκτυα που δεν είναι ανταγωνιστικά και πρέπει να συνδεθούν μεταξύ τους πιστεύουμε. Επίσης το δίκτυο ΙΤΡΙ που συνδέει την Ιταλία με την Ελλάδα και την Τουρκία είναι ένα δίκτυο το οποίο αποτελεί ένα σχέδιο σημαντικότατο. Επίσης το δίκτυο Άντρι, το οποίο συνδέει το Αζερβαϊτζάν τη Ρουμανία, το Αζερβαϊτζάν με τη Ρουμανία και με χώρες του Νότου ε, και με περιοχές και ε, περιφέρειες σε περιφερειακό επίπεδο γίνεται δηλαδή μια κατοχήρωση της ασφάλειας του εφοδιασμού. Αυτά είναι αποτελέσματα μιας κοινή ευρωπαϊκής δράσης, μιας αλληλέγγυας ευρωπαϊκής δράσης και θα μας επιτρέψει το νέο αυτό σύστημα, να, υπά, να δημιουργήσουμε ε, νέα συστήματα διασύνδεσης της Ουγγαρίας σε επίπεδο εφοδιασμού με φυσικό αέριο. Έτσι πιστεύουμε ότι πρέπει να εξετάσουμε με μεγάλη ηρεμία και μέθοδο το πώς θα χρηματοδοθούν αυτά τα σχέδια και το πώς θα γίνουν πραγματικότητα αυτές όλες οι ε, συνδέσεις για να υπάρχει μεγάλη διαφάνεια και να υπάρχει σύμφωνη γνώμη σε γενικό επίπεδο όλων των εταίρων ούτως ώστε να μπορούμε να περάσουμε στην πράξη το ταχύτερο δυνατό και να βρούμε ε, τις αντίστοιχες, τις ε, βέλτιστα προσαρμοσμένες οικονομικές λύσεις. Ένα θέμα που είναι πολύ λεπτό βέβαια. Επίσης υπάρχει και το θέμα της κατανομής του κόστους μεταξύ εθνικών κρατών και Ευρώπης. Έχουμε ανάγκη να λάβουμε μια απόφαση. Το θέμα είναι επίγον και γίνεται όλο και πιο επίγον γιατί μας πιέζει ο χρόνος και θεωρούμε ότι εμείς οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι μπορούμε να συμβάλλουμε τα μέγιστα για να υπάρξει μια διεθνική συνένεση. Γι' αυτό χαίρομαι τόσο πολύ σήμερα που δημιουργήσαμε αυτήν την κοινή εκδήλωση μεταξύ του Ουγγρικού Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να αντιμετωπίσουμε αυτό το πολύ δύσκολο πρόβλημα. Είμαι σίγουρος ότι στο πέρας της σημερινής ημέρας θα έχουμε μια ε, δυνατότητα να δούμε το πρόβλημα πιο σφαιρικά και να δούμε ε, από ποια συγκεκριμένα προβλήματα αποτελείται. Ευχαριστώ λέει ο Πρόεδρος, η κυρία Νίμπλερ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα στη σημερινή μας συνεδρίαση να απευθύνω μία άμεση έκκληση προς τους συναδέλφους από τα Εθνικά Κοινοβούλια. Έχω τρεις ε, παρατηρήσεις ε, που θα θέσω όπου υπομορφή ερωτήσεων στους συναδέλφους. Πρώτον, ε, είναι δυνατόν να έχουμε μια τέτοια ευρωπαϊκή πολιτική. το πρώτο ερώτημα σχετίζεται με την ενιαία αγορά. Είναι σαφέ ότι πρέπει να αναβαθμίσουμε τη διασυνδεσιμότητα των δικτύων μα. Αυτό είναι κάτι απαραίτητο για να δημιουργηθεί αυτή η εσωτερική Όμω Όμως ε, πολλά κράτη-μέλη συνεχίζουν να απομονώνουν τι εθνικέ ενεργειακέ του αγορέ και εφόσον οι συνάδελφοι είναι σήμερα εδώ μαζί μα, θα ήθελα να ρωτήσω, μα υποστηρίζετε, υποστηρίζετε το στόχο του ανοίγματο τη απελευθέρωση των εθνικών ενεργειακών αγορών ε, για να κατευθυνθούμε όλοι προ τη δημιουργία μέσα ενιαία αγορά Δεύτερη ερώτηση, σε σχέση με τη χρήση των ε, ανανεώσιμων πηγών ενέργεια. Ο Επίτροπο Έτιγκερ έχει εκφράσει κάποιες πολύ θαραλές ιδέες. Ε, δηλαδή άρχισε να λέει ότι ήρθε η ώρα να εξετάσουμε το ενδεχόμενο μιας ευρωπαϊκής ε, ε, αγοράς και θα πρέπει στο νότο της Ευρώπης παραδείγματος να χρησιμοποιούμε την ηλιακή ενέργεια και στο βορρά την αιωλική. Κοιτάξτε, εγώ είμαι από τη Γερμανία και όντω θα μπορούσε να είναι επαναστατική μια τέτοια κίνηση, αλλά θα ήθελα να ρωτήσω εσάς και πάλι συναδέλφους Πώς ε, νομίζετε ότι μπορείτε να προωθήσετε αυτή την ευρωπαϊκή προσέγγιση στα πλαίσια του δημοσίου διαλόγου και η Ευρώπη χρειαζόμαστε τελικά. Τρίτη ερώτηση, η Φουκουσίμα, το ατύχημα και οι επιπτώσει του. Σίγουρα στι Εθνικέ Βουλές έχετε συζητήσει με μακρόν το ζήτημα αυτό και εμεί το ίδιο και ο Επίτροπο Έτιγκερ ε, εργάστηκε πάρα πολύ σκληρά και τελικά καταλήξαμε ότι για όλες τις πυρηνικές μονάδες στην Ευρωπαϊκή Ένωση χρειαζόμαστε τεστ κόπωσης ε, και ιδιαίτερα αυστηρά κριτήρια ασφάλεια, κριτήρια συγγνώμη, ασφάλειας για όλες ε, τις πυρηνικές μονάδες ε, στην Ένωση ασχολείστε και επισταμένα με αυτό το θέμα, πιέζετε τις εθνικές σας κυβερνήσεις, ούτως ώστε να αποσκοπούν στο ε, υψηλότερο δυνατό επίπεδο ασφαλείας για όλα τα πυρηνικά εργοστάσια. Τι γίνεται με τα μέτρα ασφαλείας σε εθνικό επίπεδο. Ε, επίσης ε, θα ήθελα να συνεχίσουμε να ασκούμε πίεση για να μην επιτρέπουμε σε κανέναν να εθελοτυφλεί ε, ή να δείχνει επίοικια και χαλαρότητα σε σχέση με τις προδιαγραφές ασφαλείας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα Εθνικά Κοινοβούλια θα πρέπει να αναρωτηθούν επίσης ποια είναι η προσθέμενη αξία που μπορεί να μας προσφέρει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σας ευχαριστούμε. Από την Ιταλική Βουλή, παρακαλώ συνάδελφε, θα ήθελα εξ αρχής να σας πω ότι είναι για μένα πάρα πολύ σημαντικό να δώσω απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα της ε, κυρίας Νίμπλερ είναι ζητήματα σημαντικά όχι μόνο για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά και για τα Εθνικά Κοινοβούλια. Κυρίως για το σημερινό μας ε, ζήτημα, η περιβόητη ενεργειακή διάδρομη, θα έλεγα πρώτα απ' όλα ότι είναι σημαντικό να ε, βασιστούμε στις βασικές παραμέτρους. Τι εννοώ, η ενεργειακή διάδρομη είναι χρήσιμη για την πιο εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Αναρωτιόμαστε ή μήπως δημιουργούμε ένα νέο, μια νέα μορφή ενεργειακής εξάρτησης. Ε, σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ε, καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ούτως ώστε να... Ε, είναι λειτουργική αυτή η εσωτερική αγορά. Χάρη σε αυτούς τους λειτουργικούς όρους ε, θα υπάρξουν συγκεκριμένα ωφέλη ε, και για τους καταναλωτές και για τις επιχειρήσεις. Δηλαδή το βασικό μας κριτήριο θα πρέπει να είναι η αποτελεσματικότητα ως προς την παραγωγική δυναμικότητα, είτε μιλάμε για το πετρέλαιο είτε για το φυσικό αέριο. Και είναι καταλητικής λοιπόν σημασίας να κατοχυρώσουμε την αρχή της ουδετερότητας ε, των ε, δικτύων μεταφοράς και της διασυνδεσιμότητας, διότι οι εσωτερικές εγχώριες αγορές μπορεί να ε, πληγούν εάν δεν έχουμε ένα κρατεό ρυθμιστικό πλαίσιο, αν δεν έχουμε ε, νομική θωράκιση με αυξημένες ίσως ε, αρμοδιότητες για την για τον Οργανισμό Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αργών Ενέργειας. Χρειαζόμαστε ε, τις ε, καλύτερες τεχνικές ε, προδιαγραφές για τη λειτουργία κάθε ενεργειακής αγοράς. Ε, και μην ξεχνούμε ότι οι προσπάθειες που θα καταβάλει κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να κατευθύνονται προς αυτό το γενικότερο προσανατολισμό, δηλαδή αυτή τη δημιουργία της ενιαίας ενεργειακής αγοράς. Πιστεύω ότι για όλους μας αποτελεί προτεραιότητα το ζήτημα αυτό και ε, το μέλλον της Ευρώπης εξαρτάται από αυτό. Δηλαδή εξαρτάται από την ικανότητά μας να αντιμετωπίσουμε τέτοια ζητήματα χάρη σε μια στρατηγική θεώρηση του ε, ζητήματος και του προβλήματος αυτού. Σας ευχαριστούμε. Ο κύριος Γάινερ Βίτμα από το Αυστριακό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Το θέμα αυτό απασχολεί προφανέστατα και το Εθνικά Κοινοβούλια, πέρα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όλοι λοιπόν θα χρειαστεί να συμβάλλουν. Η κυρία Νίμπλερ αναφέρθηκε στην ηλιακή ενέργεια στον Νότο ε, και στην ε, ολική ενέργεια για το Βορρά. Ναι, ο καθένας θα κάνει ό,τι μπορεί τα δίκτυα όμως δημιουργούν μεγαλύτερη εξάρτηση. Εγώ θα ήθελα δίκτυα λειτουργικά για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θέλω να δημιουργήσουμε νέες ενεργειακές εξαρτήσεις για ορυκτά καύσιμα όπως το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο. Δεν είναι καθόλου ο επιδιωκόμενος στόχος. Ε, επίσης θα χάσουμε θέσεις εργασίας και θα χάσουμε κεφάλαια. Ε, συζητήσαμε επίσης για τη διασύνδεση των αγωγών, για τον Ναμπούκο. Το συζητάμε και στην Αυστρία. Χρειαζόμαστε τον Ναμπούκο ή όχι. Ή θα ήταν προτιμότερο να αυξήσουμε τη χρήση των ανανεώσιμων ενεργειακών πηγών. Εμεί θεωρούμε ότι, στην Αυστρία πως ε, μπορούμε να κάνουμε περισσότερα πράγματα στον τομέα τη ανανεώσιμη ενέργεια. Δεν ε, ασχοληθήκαμε καθόλου με την ενεργειακή απόδοση, με την έρευνα, με πιο θεωρητικέ ιδέε. Αλλά πέρα από αυτέ χρειαζόμαστε συγκεκριμένε προτάσει, ώστε να μα πιστέψει ο κόσμο, να μα πιστεύουν οι πολίτε Ένωση και να μπορέσουμε να κατοχυρώσουμε τον πολυπόθετο ενεργειακό εφοδιασμό. Το άλλο θέμα που μα απασχολεί είναι η ατομική ενέργεια. Εμεί έχουμε την υδροελεκτρική ενέργεια και δεν έχουμε ιδιαίτερο πρόβλημα. Ε, αλλά η Γαλλία, παράδειγμα, χάρη, έχει μεγάλη εξάρτηση από την πυρηνική ενέργεια. Ε, μακροπρόθεσμα, λοιπόν, θα έπρεπε να εγκαταλειφθεί αυτή η μορφή ενέργειας. Δεν νομίζω ότι ε, μπορεί κάποιος ε, να μιλάει με τον ίδιο τρόπο όπως το παρελθόν για την πυρηνική ενέργεια, για τα τεστ κόπωσης, ναι, το δεχόμαστε, αλλά θα πρέπει να επιτελούνται από εμπειρογνώμονες και ανεξάρτητες αρχές και όχι από τον ίδιο τον κλάδο, από την βιομηχανία. Ε, θα πρέπει να συνυπολογίσουμε και το ανθρώπινο λάθος, αλλά και τις τρομοκρατικές επιθέσεις. Εάν δεν το κάνουμε αυτό, θα ε, αφήσουμε τα λόμπι της πυρηνικής ενέργειας απλώς να κάνουν τη δουλειά τους. Δεν είναι το, το ζητούμενο. Ο στόχο δεν πρέπει να είναι μόνο η εισαγωγή ορεικτών καυσίμων από τρίτε χώρε. Θα πρέπει να βρούμε πιο καινοτόμε λύσει. Χρειαζόμαστε καλύτερη αποθήκευση επίση τη ενέργεια. αποθήκευση της ηλεκτρικής ενέργειας που προέρχεται από τις ε, συστοιχίες ε, των ε, γεννητριών όταν μιλάμε για την αιωλική ενέργεια. Επίσης το θέμα της συμπαραγωγής. Η Αυστρία έχει μεγάλη ομάδα συμφερόντων για το φυσικό αέριο. Πρέπει να συνεχίσουμε να συζητάμε για τι ανανεώσιμε πηγές ενέργειας και σταματώ εδώ γιατί δεν έχουμε χρόνο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στάνισλαν Ιβαν. Ε, εκπροσωπώ την Πολωνική Γερουσία και συγκεκριμένα την Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων. Ε, κύριοι, θα ήθελα εξ αρχής ε, να εκφράσω τη θέση της Πολωνίας από πλευράς υποδομών, ενεργειακών υποδομών και την οικοδόμηση ενεργειακών γεφύρων είναι πάρα πολύ σημαντικές. Ε, θα πρέπει να αποσκοπούμε στην ενίσχυση της ε, ενεργειακής απόδοσης. Για μας είναι ένας από τους πρωταρχικούς στόχους. Με αυτόν τον τρόπο ε, δεν θα βελτιώσουμε μόνο την κατάσταση για την ενεργειακή ασφάλεια για συγκεκριμένες χώρες, θα μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε τις αρνητικές ε, κλιματολογικές επιπτώσεις των παραδοσιακότερων ενεργειακών μορφών, συγκεκριμένα των ορεικτών καυσίμων, γιατί θα πρέπει πρώτα να ασχοληθούμε με αυτό το πρωτογενή τομέα, να το πω έτσι, και ούτω ή άλλω στο μέλλον να έχουμε περισσότερε ε, ανανεώσιμε ενεργειακέ πηγέ, τόσο το καλύτερο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα τη ενεργειακή εξάρτηση και Ακόμη σημαντικότερο είναι το θέμα της ενεργειακής απόδοσης. οφείλουμε να δημιουργήσουμε ένα χώρο καινοτομία για να προωθήσουμε τις ε, ευρωπαϊκές πολιτικές στον τομέα αυτό. Τώρα, ειδικότερα θα ήθελα να σχολιάσω ε, την κατάσταση σε κάποιες χώρες ε, και σε κάποιες περιοχές διότι όλα αυτά θα πρέπει να τα λάβουμε υπόψη, όπως είπε ο πρόεδρος Μπούζεκ, κατά την οικοδόμηση της ενιαίας ενεργειακής αγοράς. Ας πάρουμε λοιπόν την κεντρική Ευρώπη. Χρειαζόμαστε ενεργειακές γέφυρες, χρειαζόμαστε διασυνδεσιμότητα των, ενεργεια... των δικτύων. Υπάρχουν δύο συγκεκριμένα προγράμματα. Μία γέφυρα με την Λιθουανία και το δεύτερο πρόγραμμα η διασύνδεση με την Γερμανία. Πρόκειται για δύο διαφορετικές διασυνδέσεις, για να είμαι πιο συγκεκριμένος, όταν μιλάω για την Γερμανία. Και είναι απαραίτητο να λάβουμε υπόψη την σημασία της αιωλικής ενέργειας στο βορρά. Και ε, σε σχέση με τις ενεργειακές αυτές γέφυρες, θα πρέπει να εξετάσουμε με ποιο τρόπο θα βελτιώσουμε τις υφιστάμενες ενεργειακές υποδομές και πώς θα ε, δημιουργήσουμε τα FEE ε, αυτά συστήματα. Κλείνοντας, θα ήθελα να τονίσω ότι είναι απαραίτητη και η εσωτερική ε, διασυνδεσιμότητα για να αξιοποιήσουμε στο έπακρον τα συστήματα, όχι μόνο σε εθνικό αλλά και σε συνοριακό επίπεδο. Αυτό είναι απαραίτητο για την ενεργειακή ασφάλεια. Αν επιδιώκουμε τη δημιουργία ενιαίας αγοράς, αυτές ε, οι συνδέσεις ε, θα πρέπει να τύχουν τις απαιτούμενες χρηματοδότησεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε. Ζητώ συγγνώμη ε, στον γερουσιαστή. Ε, έχουμε μόνο την χώρα από την οποία προέρχεστε και δεν έχουμε την ιδιωτά σας στον κατάλογό μας, γι' αυτό και δεν την αναφέραμε. Δεν έχουμε εξάλλου μισθό τόσου πολλού βουλευτές ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σκοτσέφ. Ε, Είναι πάρα πολύ ε, σημαντικό αυτό το ζήτημα της, του ενεργειακού εφοδιασμού για τους πολίτες. Σήμερα θα περιμένατε να σας μιλήσω για την πυρηνική ενέργεια. Ε, λοιπόν, ε, όχι. Ε, θα μιλήσω για το φυσικό αέριο. Είπε ένα συνάδελφο από την Αυστρία ότι με την, σταδιακά και με τη βοήθεια των ανανεώσιμων ενεργειακών πηγών ε, θα έχουμε τη δυνατότητα να μειώσουμε την παροχή φυσικού αερίου. Δυστυχώς όλες οι αναλύσεις και εκτιμήσεις που έχω δει τουλάχιστον μέχρι στιγμής, όλες οι μελέτες λοιπόν δείχνουν πώς θα αυξηθεί η χρήση, η ζήτηση για το φυσικό αέριο στην Ευρώπη και ο βασικός λόγος, γιατί δεν θέλω να ευσέλθω σε λεπτομέρειες, ένας βασικός λόγος ε, είναι και σχετίζεται με τις ανανεώσιμες ενεργειακές πηγές έχει ως εξής. Ε, τα ενεργειακά συστήματα πρέπει να είναι ισορροπημένα και η, σταθερότητα ε, πρέπει να εξασφαλιστεί μάλλον στο συγγνώμη μια σταθερότητα ούτω ώστε να ε, αντισταθμίζουμε παραδείγματο χάρη την απώλεια ως προς το ε, παραγωγικό δυναμικό ή τα κενά στη μεταφορά της ενέργειας. Αν έχουμε όμως τέτοια προβλήματα θα χρησιμοποιούμε όλο και περισσότερο φυσικό αέριο. Άλλε πάλι χώρες θα χρησιμοποιήσουν την πυρηνική ενέργεια για να αντισταθμίσουν τις ελλείψεις ε, που παρατηρούνται σε, στην παραγωγική δυναμικότητα. Άρα στο μέλλον θα έχει ε, αυξανόμενη σημασία το φυσικό αέριο. Πώς θα τον προμηθευτούμε λοιπόν αυτό το φυσικό αέριο θα είναι ένα από τα βασικά ε, ζητήματα που θα μας αποσχολήσουν στο μέλλον. Το ο Nord Stream, ο South Stream, οι τεχνικές, ε, διασυνδε, τεχνολογικές μάλλον διασυνδέσεις με το ρωσικό δίκτυο, με αυτούς τους νέους διαδρόμους, το νότιο διάδρομο παραδείγματος χάρη μπορεί να αλλάξει άρδινη κατάσταση Ε, πρέπει όμως και να σεβαστούμε τη λογική της αγοράς. Πώς δηλαδή ε, επιθυμούμε, με ποιο τρόπο μπορούμε να δημιουργήσουμε μια πραγματική ευρωπαϊκή αγορά. Αυτό πρέπει να μας αποσχολεί και τώρα. Απευθύνω αυτό το ερώτημα στους συναδέλφους και στο πάνελ. Γιατί τα τερματικά του υγροποιημένου φυσικού αερίου ε, ασκούν τέτοια πίεση στην αγορά. Γιατί αυτή δεν χρησιμοποιούνται οι τερματικοί αυτοί σταθμοί για την ε, περαιτέρω ανάπτυξη της αγοράς και γιατί δεν ασχολούμαστε με αυτούς ε, στην στρατηγική 2020 αλλά και σε διάφορα εθνικά προγράμματα δράσης όπου υπάρχει ε, διαθέσιμη δυναμικότητα του δικτύου δοθήσεις λοιπόν τη νέα κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ρωτώ τους ε, συναδέλφου, με ποιο τρόπο ε, θα ε, βελτιώσουμε τους θερματικούς σταθμούς του υγροποιημένου φυσικού αερίου, γιατί αυτό είναι μια πραγματική ευκαιρία. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στον Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να υπογραμμίσω δύο στοιχεία που αποτελούν κλειδιά. Καταρχήν, θα ήθελα να πω ότι υπήρξε μια μελέτη ε, την οποία εκπώνησε η Ενεργειακή Επιτροπή σχετικά με την κατανάλωση της ενέργειας, της τελευταίες εβδομάδες και ε, τα απορίσματα είναι ότι έχουμε ε, τρία ε, σημεία που πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ. Το θέμα της ασφάλειας, το θέμα της κοινωνικής ασφάλειας και το θέμα της μεταφοράς των καυσίμων και ιδίω των υγροποιημένων του ευρωποιημένου φυσικού αερίου. Η Ευρώπη βεβαίως δεν αντιμετωπίζει αυτά τα θέματα με μία ενιαία φωνή. Ε, τα τελευταία δέκα χρόνια υπάρχουν πάρα πολλές συζητήσεις ε, και όλοι οι εταίροι ε, του σχεδίου South Stream άφησαν, υπέγραψαν μία κοινή συμφωνία και άφησαν τη Ρουμανία ακάλυπτη απ' έξω. Πρέπει λοιπόν να έχουμε δύο συμβόλαια. Ένα για τη μεταφορά του πετρελαίου από την Κασπία θάλασσα και επίσης ένα άλλο συμβόλαιο για τη μεταφορά του φυσικού αερίου πάλι από την Κασπία θάλασσα. Υπάρχει και το πρόβλημα του υγροποιημένου φυσικού αερίου και τελικά φτάσαμε στην περάτωση του μεγαλύτερου τερματικού για την Κορέα, την Νότια, της Ιαπωνίας και ε, το οποίο είναι η, το τέταρτο σε μέγεθος σε παγκόσμιο επίπεδο. Είμαστε λοιπόν σίγουροι ότι θα υπάρξει μια σωστή, ένα σωστός εφοδιασμός και είχαμε προβλέψει ότι θα γινόταν αυτός ο σωστός εφοδιασμός από την Κασπία θάλασσα αλλά τώρα βρισκόμαστε πάλι σε κίνδυνο γιατί υπήρξε αντικατάσταση των δυνατοτήτων παραγωγής από το φυσικό αέριο και υπήρξε και το πρόβλημα του Φουκοσίμα το οποίο άλλαξε τα δεδομένα σε παγκόσμιο επίπεδο σε ό,τι αφορά τον εφοδιασμό της ενέργειας 72 μονάδες ε, ε, πυρηνικής ε, ενέργειας προβλεπόντουσαν. Δεν είμαστε σίγουροι ε, γιατί τα τελευταία χρόνια ε, οικοδομήθηκαν μόνο εννέα τέτοιες πυρηνικές μονάδες. Υπήρχε δηλαδή μεγάλη αισιοδοξία σε σχέση με τις τα προγράμματα αυτά. χρειάζεται όμως να καταλάβουμε ότι αυξήθηκε η κατανάλωση τα τελευταία χρόνια ε, σε υγρά καύσιμα και ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας το επιβεβαιώνει αυτό και επίσης ένας οργανισμός ο οποίος μιλάει για το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ενέργειας στον Καναδά διαπιστώνει ότι ε, θα αυξάνονται συνέχεια ε, και θα αυξηθούν περαιτέρω τα υγρά καύσιμα και κατανάλωσή τους κατά με ένα ποσοστό 81% στα επόμενα 10 χρόνια δεν έχουμε μόνο ένα στοιχείο για τα υγρά καύσιμα. Πρέπει να ξέρουμε α, τι διαθέτουμε. Έχουμε μια αγορά ε, φυσικού αερίου. Σωστή. Ε, είναι, είμαστε πάρα πολύ αισιόδοξοι όταν λέμε ότι θα έχουμε περατώσει μια ενιαία αγορά σε φυσικό αέριο μέσα σε τέσσερα χρόνια για το φυσικό αέριο είναι αδύνατο. Μπορεί να είναι δυνατό για το πετρέλαιο, δεν ξέρω. Σας δίνω το παράδειγμα της Ρουμανίας, όπου στη Ρουμανία η οποία βρίσκεται στα όρια του ευρωπαϊκού χώρου και εξαρτάται από μια ενιαία πηγή, δηλαδή τη Ρωσία, δεν έχουμε εμεί αγορά φυσικού αερίου. Λοιπόν, η αύξηση της εξάρτησής μας από τις εισαγωγές από την Ευρωπαϊκή Ένωση καθιστά αδύνατη τη δημιουργία μιας αγοράς, μιας πραγματικής αγοράς με την πραγματική σημασία του όρου και πρέπει να κατανοήσουμε ότι η πρόταση να δημιουργηθεί μια επιτροπή ενέργειας σε επίπεδο κρατών μελών είναι κάτι των εξών κάνευ. Χρειάζεται επίσης μια στρατηγική ευρωπαϊκών συμφερόντων και επίσης πηγές χρηματοδότησης, να μπορεί να υπάρξει εγγύηση ετήσιας χρηματοδότησης η οποία να έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα για το καθένα από αυτά τα σχέδια. Διότι διαφορετικά ε, θα παραμείνουμε στις γενικές συζητήσεις. Δεν θα μπορέσουμε να περάσουμε σε πράξη. Έχουμε πολλά κράτη βεβαίως που πέρασαν την κρίση και εφόσον την πέρασαν τώρα ε, μιλάν μόνο ε, με ε, εθνικιστικές βλέψεις. Ε, θα ήθελα να πάψει να υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι το ενεργειακό. Η ενέργεια γίνεται όλο και ακριβότητη και στο οικονομικό περιβάλλον και στο κοινωνικό. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να γίνει στρατηγική προτεραιότητα η ενέργεια σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. περνάει η ώρα πολύ πιο γρήγορα από ό,τι προβλέψαμε. Πέρα από τα τρία άτομα τα οποία είναι γεγραμμένα ε, στον πίνακα ή στην οθόνη ε, θα πρέπει να περατώσουμε. Έχουμε τη σύνθεση της συζήτησης ε, στο τέλος. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Σούλτες του Ευστριακού Κοινοβουλίου. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ που μου δώσατε το λόγο. Αξιότιμοι συνάδελφοι, πρόκειται για τη μείωση ε, των ε, ε, εκπομπών διοξιδίου του άνθρακος και για τη δημιουργία διαδρόμων. Καταρχήν για το φυσικό αέριο. Το φυσικό αέριο ήταν ένα θέμα που, για το οποίο συζητήθηκε πάρα πολύ το θέμα της αποτελεσματικότητάς του. Στην Αυστρία το 90% του φυσικού αερίου περνάει από την επικράτεια και η μεταφορά αυτή ε, γίνεται με πολύ μεγάλες εκπομπές 500.000 ε, τόνων διοξιδίου του άνθρακος όπως καταμετρήθηκε πρόσφατα ε, και θα πρέπει να αυτές οι οδικές μεταφορές να κατανοήσουμε ότι είναι πάρα πολύ επιβλαβείς ε, και δεν ξέρουμε πώς θα δημιουργηθεί αυτός ο ενεργειακός διάδρομος, τι αποτελεσματικότητα θα έχει. Πρέπει να βελτιωθεί ε, η μεταφορά του φυσικού αερίου οπωσδήποτε και βεβαίω αυτό το γράφει το σημερινό κείμενο και να υπάρχει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα για την κατασκευή του ηλεκτρικού ρεύματος αλλά το ίδια η μεταφορά έχει πρόβλημα. Δεν είναι αποτελεσματική η μεταφορά φυσικού αερίου. Γι' αυτό θα πρέπει στις ε, περαιτέρω διαβουλεύσεις το στοιχείο αυτό να ληφθεί σοβαρά υπόψη. Τώρα, το θέμα του ηλεκτρικού ρεύματο, Εμείς στην Αυστρία πιστεύουμε ότι το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό όχι μόνο ως πολιτική συζήτηση αλλά και ως ανησυχία του πληθυσμού Πιστεύουμε ότι ε, το διαμετακομιστικό εμπόριο που γίνεται μέσα από την Αυστρία ε, έχει πάρα πολλές συνέπειες και θέλουμε να ξέρουμε από πού προέρχεται το ηλεκτρικό ρεύμα και κατά πόσο οι, πυρηνικοί, οι πυρηνικές εγκαταστάσεις που παράγουν ηλεκτρικό ρεύμα έχουν μεγάλη σημασία. Για να γίνει αποδεκτό το σχέδιο αυτό από τον πληθυσμό ενδεχομένως σε γενικές γραμμές πρέπει να αναρωτηθούμε πιστεύω εάν αυτή η μεγάλη ενεργειακή διαδρομή είναι το μόνο θέμα το οποίο ε, πρέπει να συζητήσουμε την παρούσα στιγμή γιατί προσφέρει μια περιφερειακή δομή. Αυτή η περιφερειακή δομή ε, θα είναι πολύ σημαντική για τα δίκτυα της, ε, του ελάχιστου εφοδιασμού για να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε διάφορες εναλλακτικές πηγές ενέργειας, ανανεώσιμες, τη βιομάζα κτλ. Θα πρέπει να ε, είναι διαθέσιμες αυτές οι πηγές και γιατί υπάρχουν αυτοί οι μεγάλοι διάδρομοι, αλλά το θέμα είναι ευαίσθητο. Για τους μεγάλους διαδρόμους ε, έχουμε συζητήσει κατά επανάληψη και θεωρήσαμε ότι είναι πάρα πολύ ακριβή, ότι οι χώρες προέλευσης αρνούνται να καταβάλουν αυτά τα τεράστια ποσά και πρέπει να, κατα... να λάβουμε υπόψη μας ότι ο κάθε μεγάλος ενεργειακός διάδρομος μας κάνει να χάνουμε σε ευρωπαϊκή αξία. θα πρέπει να ενισχύσουμε την αποδετικότητα, να έχουμε μια πραγματική διαφοροποίηση στην προέλευση την ενεργειακή. Υποστηρίζω πλήρως το θέμα του υγροποιημένου φυσικού αερίου που θα μπορούσε να μεταφερθεί ε, με πλοία. Τα τερματικά είναι απαραίτητα και θα πρέπει να αποτελούν μια πραγματική εναλλακτική λύση. Κάτι το σημαντικό, αν εισάγουμε φυσικό αέριο θα πρέπει να ξέρουμε ότι πάρα πολλές χώρες από όπου προέρχεται το αέριο δεν είναι δημοκρατικές χώρες. Δεν ξέρω αν τις θεωρούμε ως δημοκρατίες, αλλά πάντως ξέρουμε ότι ότι στέλνοντας χρήματα σε αυτές τις χώρες δεν υποστηρίζουμε, τις, τη σταθερότητα αυτές τις χώρες αλλά τα ολοκληρωτικά καθεστώτα. Αν παραδείγματος χάρη πρόκειται για το Ιράν δεν μπορούμε να είμαστε υπερήφανοι όταν στέλνουμε εκεί τα χρήματά μας. Ποια είναι η σταθερότητα του εφοδιασμού ε, με τον Αμπούκο θα έπρεπε να λειτουργήσει αλλά δεν υπάρχει εμπιστοσύνη εκ μέρους των επενδυτών σε σχέση με την ασφάλεια του αερίου. Ιδαλλιώ θα είχε κατασκευαστεί εδώ και πάρα πολύ καιρό. Δεν μπορούμε να δώσουμε απάντηση στο θέμα αυτό. Λέμε ακόμα ένα χρόνο, ακόμα ένα χρόνο, ακόμα ένα χρόνο, αλλά δεν έχουμε ακόμη απαντήσεις. Και αν διαρωτηθούμε... αν δεν θα υπάρξουν μεγάλα έργα με μεγάλους διαδρόμους, με μεγάλη χωρητικότητα που συζητούνται. Αλλά θα ήθελα να σας πω ότι η πιο ασφαλής ενέργεια δεν είναι αυτή που μεταφέρεται σε μεγάλη κλίμακα, αλλά αυτή που μπορούμε να έχουμε πολύ πιο εύκολα. Διότι με την αύξηση της αποδοτικότητας και καλύτερη χρήση αυτής της ενέργειας μπορούμε να επιτύχουμε καλά. Πώς η Ευρώπη χρειαζόμαστε, αυτό είναι πάρα πολύ εύστοχο ερώτημα. Αυτή τη στιγμή με την αντίληψη των οικονομιών μας πρόκειται για μακροπρόθεσμα συμβόλαια και αυτό συνδέει την δυναμικότητα των δικτύων και δεν υπάρχει ανταγωνισμός και θα ήθελα να ζητήσω από τα ευρωπαϊκά όργανα να προσπαθήσουν να ξαναεξετάσουν αυτή τη διάσταση. Και ένα σίγουρο πράγμα, η Ευρώπη γεννήθηκε μετά από τα θέματα που βασιζόντουσαν στον άνθρακα και στον χάλιβα. Και τώρα έχουμε τη σημερινή κρίση, ίσως είναι απαραίτητο τα θέματα τα ενεργειακά να θεωρηθούν ένα θέμα ευρωπαϊκό να συζητήσουμε μαζί και να λάβουμε γρήγορα αποφάσεις για να προχωρήσουν τα πράγματα. Ευχαριστώ πολύ. Άντρας Γιώργη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ πολύ. έχετε εξαγάγει συμπεράσματα. Θα ήθελα να αντιδράσω ε, εντάχει στα όσα ακούσαμε μέχρι τώρα. Υπάρχουν πολλοί βουλευτές ε, που έλαβαν ε, το λόγο για το μείγμα το ενεργειακό και το θέμα της πυρηνικής ενέργειας. Και σύμφωνα με τις διάφορες παρεμβάσεις νομίζω ότι πιστεύουμε σε μια ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας, χρειαζόμαστε μια εσωτερική αγορά ενέργειας και αυτό θα είναι προς όφελος όλων. Αλλά θα υπάρξουν πάντοτε ε, θέματα, τομείς που να εξαρτώνται από τα κράτη-μέλη λόγω της αρχής της επικουρικότητας. Αυτό είναι προφανές, αλλά είναι σημαντικό να κάνουμε διάκριση ανάμεσα στις κοινέ αρμοδιότητες και στις αρμοδιότητες των κρατών μελών. Αυτό είναι προφανές. Μια κοινή εσωτερική αγορά θα ήταν κάτι το κοινό, μια κοινή αρμοδιότητα. Και αυτό το βλέπουμε, το βρίσκουμε στο τρίτο πακέτο ενέργειας και είναι σαφές ότι η δημιουργία των απαιτουμένων υποδομών για αυτήν την αγορά ενέργειας είναι σημαντικές. Γι' αυτό ασχολούμεθα με τους ενεργειακούς διαδρόμους σήμερα και είναι ο λόγος για τον οποίο υιοθετούμε τις νομοθετικές πράξεις που επιτρέπουν την ενεργειακό εφοδιασμό. Αυτό το μείγμα το ενεργειακό είναι αποφασιστικό, διότι οι καλύτερες αποφάσεις στον τομέα αυτό θα μπορούσαν να ληφθούν σε επίπεδο εθνικό και περιφερειακό. Αυτό ισχύει και για το θέμα των εναλλακτικών ε, πηγών ενέργειας. Αυτό εξαρτάται από τα κράτη-μέλη και είναι σαφές ότι το ενεργειακό μείγμα είναι στο τομέας αρμοδιότητας και στο επίπεδο το πυρηνικό και εκεί πρέπει η απόφαση να ληφθεί σε εθνικό επίπεδο. Όταν εδώ στις Βρυξέλλες μιλούμε για το θέμα αυτό, όταν βλέπουμε ποιες είναι οι συνέπειες του ατυχήματος στη Φουκουσίμα όλοι θα θυγούμε και θέλουμε όλοι να λάβουμε το λόγο και όταν μιλούμε για ασφάλεια πρόκειται για κάτι το οποίο, στο οποίο αποδίδεται ιδιαίτερη σημασία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και όσον αφορά στο ενεργειακό μείγμα και στο ενεργειακό μείγμα για το μέλλον πρέπει ε, να είμαστε ήρεμοι. Δεν χρειάζεται γρήγορα γρήγορα ε, εντάχει να λάβουμε αποφάσεις ε, βιαστικές. Πρέπει να επιδείξουμε αλληλεγγύη και είναι ο λόγος για τον οποίο η Ουγγρική Προεδρία αντέδρασε με αποτελεσματικότητα, με ταχύτητα, αλλά πρόκειται για κάτι που είναι της αρμοδιότητας των κρατών μερών. Από την άλλη πλευρά, αν θέλουμε μια ενιαία ευρωπαϊκή αγορά, μια ενιαία ευρωπαϊκή πολιτική, θα πρέπει να είμαστε σαφείς για τους τομείς της εθνικής αρμοδιότητας και τους τομείς ευρωπαϊκής. Ο πρόεδρος, ο κύριος από το Κοινοβούλιο του Λουξεμβούργου. Ευχαριστώ. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να επιστήσω την προσοχή σας σε ένα σημείο. Ο τρίτος άξονας της στρατηγικής 2020, δηλαδή το 20% σε σχέση με την ενεργειακή απόδοση, νομίζω ότι θα πρέπει σήμερα εδώ να συζητήσουμε και αυτό το θέμα, διότι δεν ε, πρέπει να ε, παράγουμε ενέργεια για την ε, καταναλώνουμε άσκοπα στη συνέχεια. Πέρα από την κατασπατάληση της ενέργειας, ε, παραβλέψαμε ε, και διάφορα άλλα σημαντικά ζητήματα. Μιλήσατε για τους ενεργειακούς διαδρόμους, αλλά ε, η Γαλλία και η Γερμανία από τις χώρες Μπενελίξ έχουν ιδρύσει ένα φόρουμ πέντε κρατών με, με κοινή διάθεση ενεργειακών πόρων πέρα από τα σύνορα των χωρών αυτών. Ε, η υπεράκτια, παραδείγματο χάρη, η ενέργεια από τη βόρεια θάλασσα μπορεί να εισαχθεί και το Λουξεμβούργο, μια μικρή χώρα, είχε την πρόθεση να προσφέρει για την αποθήκευση 11.000 ε, ΜΒ τι εννοώ, γίνεται μια ενδιάμεση αποθήκευση κατά τη μεταφορά της ενέργειας και θα παρουσίαζε ιδιαίτερο ενδιαφέρον αν έκαναν ακριβώς το ίδιο και μεγαλύτερες χώρες, ε, δηλαδή αν ε, κατασκεύαζαν τέτοιες ε, μονάδες ενδιαμέσου αποθήκευσης. Ε, πέρα από την Αυστρία θα μπορούσαν χώρες όπως η Δανία και το Ηνωμένο Βασίλειο αλλά και η Νορβηγία να κάνουν παρόμοιες κινήσεις διότι και η Νορβηγία μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτές τις μονάδες αποθήκευσης. Λοιπόν, μιλώντας για την ενεργειακή αγορά θα πρέπει να τονώσουμε αυτή την αγορά με τέτοιες κινήσεις. Δεύτερον, ε, είπαμε ότι δεν είναι ευταίο να εξαρτώμεθα από χώρε όπω η Ρωσία για τον ενεργειακό μα εφοδιασμό ή από χώρε ε, τη Μέση Ανατολή, είτε μιλάμε για το πετρέλαιο είτε για το φυσικό ε, αέριο. Δεν πρέπει να ξεχνάμε προγράμματα όπως το πρόγραμμα συνεργασίας με τις χώρες του Μαγκρέμπ. Τώρα βέβαια με την Αραβική Άνοιξη δεν ήρθε η κατάλληλη στιγμή για να γεννηθεί αυτό το πρόγραμμα Mare Nostrum που είχαμε προγραμματίσει. Έτσι θα γίνει και καλύτερη χρήση του προγράμματος Serimu Desert. Σε έξι ώρες ο ήλιος μπορεί να μας δώσει ε, την ενέργεια που χρειάζεται για μια ολόκληρη ημέρα γη. Νομίζω ότι θα έπρεπε να διατηρήσουμε επαφές με τις χώρες του Μαγκρέπ, παρότι έτσι δημιουργούμε μια νέα εξάρτηση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Οι τελευταίες παρεμβάσεις θα ακολουθήσουν τώρα. Από, πρώτα απ' όλα από έναν βουλευτή του Ουγγρικού Κοινοβουλίου. Είδαμε με ποιο τρόπο Ε, ε, κάποιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, δεν δεσμεύτηκαν για τους ενεργειακούς διαδρόμους που σχεδιάζουμε σε επίπεδο ένωσης, σε περιφερειακό επίπεδο, έκαναν επενδύσεις αλλά ασχολήθηκαν με τον δικό τους εφοδιασμό και μόνο. άρα δεν μπορούμε να επιδιώκουμε μέσω πρόθεσμα μείωση των τιμών αν συνεχίσουμε έτσι. Υπάρχουν πολλές αντιφάσεις προς το παρόν. Πρώτα απ' όλα, σε σχέση με την κρίση διαπιστώσαμε ότι ε, διαρκώς αυξάνουν τα κράτη-μέλη τους ενεργειακούς φόρους. Αυτό δημιουργεί μεγαλύτερη ανασφάλεια ε, ως προς τις επενδύσεις ε, στον κλάδο. Ε, επίσης, ε, υπονομεύει τη διαφάνεια στην ενεργειακή αγορά. Αυτό τι σημαίνει ότι οι μεγάλες επενδύσεις που απαιτούνται για την δημιουργία αυτών των ενεργειακών διαδρόμων δεν θα είναι βιώσιμες για τις επιχειρήσεις. Ως εκ τούτου, πολύ συχνά δεν γίνονται οι επενδύσεις διότι θεωρήθηκε ότι εν λόγω εταιρείες δεν θα είναι αρκετά κερδοφόρες ε, ή ότι δεν θα είναι γρήγορα κερδοφόρες. Νομίζω ότι ε, ο στόχος μας θα πρέπει να είναι να εκπονήσουμε μία νέα μέθοδο, ούτω ώστε να συνεργαστεί η βιομηχανία με το κράτος για τα ενεργειακά ζητήματα. Θα πάρω ένα ε, παράδειγμα από τη δική μου χώρα. Βλέπουμε πως η συνεργασία που βασίζεται σε ενιαίες αρχές βασίζεται σε συνεργασία ερευνητών ε, και εταιριών. Μπορούμε δηλαδή να αναπτύξουμε τέτοιες λύσεις, ούτως ώστε να συνεργάζονται καλύτερα τα ερευνητικά ιδρύματα, αλλά και οι βιομηχανίες. Τώρα, ένα άλλο θέμα είναι αυτό των εξαγωγικών βιομηχανιών ε, κάποιων ε, κρατών Ε, δεν θα πρέπει να παραγνωρίσουμε τη σημασία του κεφαλαίου. Οι εταιρείε που διαθέτουν το κεφάλαιο για την έρευνα επηρεάζουν και τις εξελίξεις. Και το θέμα είναι ότι ε, οι εταιρείε που δραστηριοποιούνται στον ε, κλάδο αυτό μπορεί να είναι λιγότερο ή περισσότερο κερδοφόρε. Οπότε θα πρέπει να εξετάσουμε ταυτόχρονα και του κανόνε για τι κρατικέ επιδοτήσει για το προσδιορισμό των τιμών, των, του, τους κανόνες που θα ισχύουν για τις τιμές, νομίζω ότι είναι καλύτερο να παρέμβουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο και όχι σε εθνικό. Σας ευχαριστούμε. Παρακαλώ, έχετε ζητήσει το λόγο. Εκτός μικροφώνου δεν ακούνε διερμηνείς, δυστυχώς. Δεν θα συνοψίσω. Θα ήθελα να κάνω κάποιες σύντομες παρατηρήσεις σε σχέση με αυτές ε, τις τόσο εύστοχες και ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις που έκαναν οι βουλευτές. Η ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική συγκεκριμένα είναι συνδυασμός αυτών που γίνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε εθνικό επίπεδο αφετέρου. Πρέπει να είναι αλληλοσυμπληρούμενες αυτές οι δράσεις και βεβαίως να λαμβάνεται υπόψη το νομικό σύστημα. Να δούμε δηλαδή αν η νομική κατάσταση δικαιολογεί την παρέμβασή μας σε επίπεδο ένωσης. Ε, βέβαια δεν είναι αυτός σκοπός, είναι λογικό να γίνουν πιο ανταγωνιστικές οι αγορές, να είναι ασφαλέστερος ο εφοδιασμός των μεμονωμένων κρατών και των εταιριών. Θα ήθελα να κάνω μια διάκριση, μια διευκρίνηση. Η εξάρτηση της ενεργειακής αγοράς ε, τι σημαίνει. Εξάρτηση μέσα σε ένα ένομο σύστημα, δηλαδή κατοχυρώνεται η αλληλεξάρτηση μέσα από το νομικό σύστημα. Η εξάρτηση σε σχέση τώρα με τις τρίτες χώρες ε, είναι κινούμενοι άμμος, γιατί ε, ισχύουν διαφορετικά συστήματα. Εάν τώρα μιλάμε για την διασύνδεση ανάμεσα στην Αυστρία και την Ιταλία, αν πιστεύουμε ότι είναι πρόσφορο, έτσι, εγώ πιστεύω ότι είναι, γιατί θα υποφεληθούν οι Ιταλικοί, οι Ιταλοί, συγγνώμη, καταναλωτές και οι Ιταλικές εταιρείε. Αυτό προβλέπεται από την νομοθεσία και το ίδιο ισχύει εξάλλου και για την αποθήκευση αλλά και για την πυρηνική ασφάλεια. Γιατί είναι τόσο σημαντικό αυτό το θέμα για τον Επίτροπο Έτιγκερ και γενικότερα για την Επιτροπή, διότι χώρε που δεν έχουν πυρηνική ενέργεια ανησυχούν για τις επιπτώσεις αυτή τη βιομηχανία. Οι χώρε που ε, δεν έχουν ε, μονάδε θέλουν παρόλα αυτά να εφαρμόζονται οι ύψιστε προδιαγραφέ ασφαλεία και γι' αυτό χρειάζεται. Ε, χρειάζονται, χρειάζονται συνδυασμένε προσπάθειε για να τα καταφέρουμε σε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Υπάρχει ένα ε, τομέα όπου δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα, αλλά μπορούμε να λάβουμε δράση για την πρόληψη των τρομοκρατικών χτυπημάτων, γιατί πρόκειται για εθνική αρμοδιότητα. Φυσικά δεν μπορούμε να ελέγξουμε εμεί ε, την MI6 του Λονδίνου ή την Υπηρεσία Πληροφοριών τη Γερμανία από τι Βρυξέλλε, αλλά μπορούμε να ασχοληθούμε με τι ελλείψει στην ασφάλεια λόγω τρομοκρατικών χτυπημάτων. Αυτό εμπίπτει στην αρμοδιότητά μα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους βουλευτές και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και από τα Εθνικά Κοινοβούλια, διότι ε, σχολίασαν διάφορες διαστάσεις του ζητήματος που πρέπει να συνυπολογίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρωτού καταθέσει την επίσημη πρότασή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς σας ευχαριστούμε και τώρα για τη σύνοψη ο κύριος Σορότσκι έχει τον λόγο. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Υπουργέ. Θα ήθελα να αρχίσω την ε, παρέμβασή μου κάνοντας ε, ένα προσωπικό σχόλιο. Πρώτη φορά έρχομαι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και βρίσκω ότι είναι καταπληκτικό αυτό που συμβαίνει εδώ σήμερα. Συμφωνούμε μεν για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά διαπιστώνουμε ότι ε, διείστανται απόψεις για πολλά ζητήματα. Βεβαίως ε, είναι πολύ ενδιαφέρουσες αυτές οι διαφορετικές απόψεις. Ε, κατά την εξέβρεση συνένεση λοιπόν θα πρέπει να ασχοληθούμε με κάποια βασικά ζητήματα. Συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αναλάβει δράση για να κατοχυρώσει τον ενεργειακό εφοδιασμό και χρειάζεται μια κοινή ενεργειακή πολιτική. Αυτό θα λειτουργήσει ως εφαλτήριο που θα μας επιτρέψει να συνεχίσουμε τις προσπαθίες μας. Βεβαίως θα πρέπει να έχουμε συμφωνήσει επί αυτό το σημείο πριν μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Προκύπτει σαφέστατα από τον σημερινό μας διάλογο ότι οι υφιστάμενες υποδομές, ο εξοπλισμός είναι, ε, αν θέλετε, μια κοινή, ένα κοινό αγαθό για όλα τα κράτη-μέλη. Ε, μέχρι στιγμής ασχολούμασταν με τσογούς με μεταφοράς πετρελαίου και την διασύνδεσή τους. Ένας αυστριακός βουλευτής μίλησε επίσης και για τα ε, δίκτυα ηλεκτρικής ε, ενέργειας ε, και για τα προβλήματα που δημιουργούνται διότι δεν επιθυμούν οι αυστριακοί καταναλωτές ηλεκτρική ενέργεια που να έχει παραχθεί σε πυρηνικό εργοστάσιο. Εν γέννη βέβαια δεν διαπιστώνουν ότι υπάρχουν σοβαρά προβλήματα για την διασυνδεσιμότητα των ηλεκτρικών δικτύων για την διασυνδεσιμότητα τώρα των αγωγών φυσικού αερίου. Αυτό σαφέστατα θα έχει μεγάλες επιπτώσεις επί της ενεργειακής ασφάλειας, ασφάλειας ανεφοδιασμού ε, και την εσωτερική αγορά ενέργειας. Ακούσαμε πολύ άριθμα σχόλια ενδιαφέροντα που με ποιους τρόπους παραδείγματος χάρη μπορούμε να περιστήλουμε την ενεργειακή μας εξάρτηση και ένας συνάδελφος από το Λουξεμβούργο εξέφρασε την, το, το όραμα του που εφαρμόζεται ήδη στις ε, χώρες ε, Μπενελούξ και λειτουργεί ε, ομαλά η αγορά χάρη σε αυτή την κοινή δράση. Να λοιπόν ένα λαμπρό παράδειγμα για τις μελλοντικέ μας δράσεις. Θα έπρεπε λοιπόν να διευρύνουμε τέτοιου είδους επιτυχημένα προγράμματα σε ολόκληρη την επικράτεια της Ένωσης. Ε, πολλοί συνάδελφοι μίλησαν για τις μελλοντικέ προκλήσεις, ε, για τη δυνατότητα που έχουμε να βρούμε συγκεκριμένες λύσεις. Για ένα σημείο διαπίστωσα ότι υπάρχει συμφωνία. Ε, πιο συγκεκριμένα το θέμα της ενεργειακής εξάρτησης ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, έχει ως αποτέλεσμα να είμαστε σε ασθενή διαπραγματευτική θέση για τα ενεργειακά ζητήματα σε παγκόσμιο επίπεδο. Ακούσαμε επίσης ότι ως πολιτικοί δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε δράσεις και προγράμματα σε συνεργασία με χώρες που δεν θεωρούμε δημοκρατικές ε, τα έσχατα γεγονότα στη Βόρεια Αφρική ευτυχώς έδειξαν ότι ε, δεν ε, είναι παντοτινές οι δικτατορίες Βεβαίω, ε, παρατηρούμε ταυτόχρονα ότι χρειάζεται αποτελεσματική εξωτερική πολιτική για την Ένωση αν ε, προτίθεται να έχει αποτελεσματική ε, ενεργειακή πολιτική. Άλλο θέμα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε είναι αυτό της πυρηνική ενέργειας όπως είπαν πολλοί συνάδελφοι και ε, φαίνεται ότι συμφωνούμε ε, σχετικά με τα τεστ κοπόσεως που εισηγήθηκε ο Επίτροπος Έτιγκερ. Φαίνεται να συμφωνείτε ότι πρέπει να διεξαχθούν ε, οι έλεγχοι αυτοί. Είπανε κάποιοι βεβαίως ότι τα τεστ θα πρέπει να διεξαγάγονται από πυρογνώμονες ή ανεξάρτητες αρχές. Θα αναμείνουμε προς το παρόν τη σχετική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ταυτόχρονα στην πράξη ε, καλούμαστε να λάβουμε αποφάσεις ε, για τις προδιαγραφές διεξαγωγής ε, των τεστ κοπόσεως. Ο προβληματισμός θα είναι συλλογικός και για την ενεργειακή ασφάλεια, πέρα από το να είμαστε ανταγωνιστικοί, χρειαζόμαστε και τη συνεργασία και την αλληλεγγύη. Φαίνεται όμως ότι υπάρχει αυτή η πολιτική βούληση ε, για να υπάρξει έμπρακτα η ενεργειακή αλληλεγγύη και φαίνεται ότι υπάρχει επίσης κοινή βούληση για να κατευθυνθούμε προς μια κοινή ενεργειακή πολιτική στην Ένωση μελλοντικά. Ε, πλην όμως δεν θα πρέπει να λησμονήσουμε πως ε, ε, όλες αυτές οι προτάσεις έχουν επιπτώσει ως προς τη χρηματοδότηση και τον προϋπολογισμό και όλα αυτά θα ε, πρέπει να τα έχουμε κατά νου όταν ε, συντάσσουμε τους νέους κανονισμούς. Επίσης έχει σημασία αυτό για την εφαρμογή των προγραμμάτων. Ή, οφείλουμε να σκεφτούμε και τα συμφέροντα των επενδυτών. Η κερδοφορία τέτοιων ε, προγραμμάτων ε, έχει κέριο ρόλο. Επίσης ε, θα περιμένουμε από τα νοικοκυριά και τους καταναλωτές να συμβάλλουν σε αυτή τη συλλογική προσπάθεια. Όλοι θα πρέπει να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες της ενιαίας αγοράς και ξαναλέω ότι θα πρέπει να μελετήσουμε ενδελεχώς το ζήτημα προτού καταθέσουμε νέες προτάσεις. Άλλο θέμα τώρα, εναρμόνιση των τεχνικών προδιαγραφών. Εγώ συμφωνώ πως χρειαζόμαστε μία διαδικασία ενιαίας αδειοδότησης για τους ενεργειακούς ε, διαδρόμους. Όμως, ε, προς το παρόν, οι εθνικές αρχές ε, κατέχουν την αρμοδιότητα για αυτό το θέμα. Ιδού, αυτό. Αυτά ήταν τα σημεία που μας απασχόλησαν σήμερα και πιστεύω ότι ε, μέσα από το διάλογο ε, σφυριλατούμε τις μελλοντικέ κοινέ μας ε, θέσεις. Διάφοροι συνάδελφοι, μεταξύ των οποίων και ο Γερμανός συνάδελφος, ξεκαθάρισαν ότι στα εθνικά μας κοινοβούλια πρέπει να προαγάγουμε την περαιτέρω την ευρωπαϊκή διάσταση της ενεργειακής πολιτικής, ε, να παραμερίσουμε τα εθνικά μας ε, συμφέροντα, ούτως ώστε να συνεργαστούμε όλοι για την πρόθεση των ευρωπαϊκών συμφερόντων. Πιστεύω ότι όλα τα μέλη του Ιγκουρικού Κοινοβουλίου θα συμφωνήσουν και θα ακολουθήσουν αυτή την κατευθυντήρια αρχή στις μελλοντικέ τους εργασίες. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ όλους τους μετέχοντες ε, για τις παρεμβάσεις τους και τώρα ο κύριος ε, Ρόιλ θα προεδρεύσει στο επόμενο τμήμα της συζήτησής μας και του δίνω το λόγο. Αγαπητοί συνάδελφοι, ε, περνάει ο χρόνος και διαπιστώνω με δέος ότι ξεπεράσαμε το χρόνο που είχαμε στη διάθεσή μας και διαρωτώ με εάν δεν πρέπει να συνεχίσουμε ε, με το δεύτερο μέρος χωρίς να κάνουμε μεγάλο διάλειμμα. Ιδαλλιώς δεν θα έχουμε χρόνο. Αν συμφωνείτε θα μπορούσαμε να μην κάνουμε διάλειμμα και να αρχίσουμε τη συζήτηση. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει ίσως να προβλέψουμε τρία λεπτά για κάθε παρέμβαση, αλλά μέχρι τώρα δεν έχει ζητήσει κανείς τον λόγο αυτό μου περιπλέκει το έργο μου ή μου το διευκολύνει. Δεν ξέρω πώς θα το εκλάβετε αυτό. Α, είδαμε κάποιον που θέλει να λάβει το λόγο. Ο πρώτος που εκδηλώθηκε είναι λίγο δύσκολο. Α, ναι. Ναι. Κυρία Χέρτσοκ, είσαστε παρούσα. Θα αρχίσουμε με αυτό, αν συμφωνείτε. Θα ήθελα τώρα, αν συμφωνείτε, θα ήθελα να δώσω το λόγο στην εισηγήτρια την κυρία Χέρτσοκ. Η κυρία Χέρτσοκ πρώτα απ' όλα. Thank you, thank you, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Παρόλο που είμαι από την Ουγγαρία αποφάσισα να μιλήσω αγγλικά διότι θα ήθελα να δείξω ότι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έχουμε εθνικές σημαίες, έχουμε πολιτικές σημαίες. Εγώ ανήκω στο Σοσιαλιστικό Κόμμα και εργάζομαι για θέματα που σχετίζονται με την ενέργεια. Αλλά στις 5.30 θα πρέπει ακριβώς να φύγω γιατί έχουμε είμαι σκιώδης εισηγήτρια για ένα θέμα πυρηνικής ενέργειας. Δεν μπορώ να μείνω πέραν των 5.30 αλλά θα κάνω ό,τι μπορώ για να καλύψει το θέμα. Αλλά δυστυχώς ε, το καθήκον με καλή και είναι πολύ σημαντικό αυτό το καθήκον. Γιατί πρέπει να σας μιλήσω. Όταν μιλούμε για τις ενεργειακές πολιτικές νομίζουμε ότι πρόκειται για πόρους ενεργειακούς, ε, για οδούς διέλευσης, ε, για ενεργειακή τεχνολογία κλπ. Και Πάρα πολύ συχνά πιστεύουμε ότι η ενεργειακή πολιτική είναι όλα όσα έχουν συζητηθεί στην προηγούμενη συζήτηση. Αλλά όταν μιλούμε για ενεργειακή πολιτική έχουμε το δεύτερο τμήμα, το δεύτερο μέρος της συζήτησης όταν η ενέργεια φτάνει στους καταναλωτές και αυτό είναι εξίσου σημαντικό όπως η προηγούμενη συζήτηση και πρέπει να γίνουν πάρα πολλά πράγματα όπως και για το προηγούμενο θέμα. Όταν ήρθα πριν από 7 χρόνια στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήταν για πολλούς έκπληξη ότι μια γυναίκα ενδιαφέρεται για τα ενεργειακά θέματα. Μου είπαν ότι τα θέματα ενέργειας είναι περισσότερο για τους άνδρες. Ε, τότε υπήρχε επίτροπος ε, που πίστευε ότι έχει και ανθρώπινη μορφή ενέργεια και αφορά ε, τις γυναίκες. Αυτό το σκεφτόταν ο Επίτροπος ε, Πίμπαλξ ε, αλλά αφορά όμως όλη την Ευρώπη και τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά. Νομίζω ότι το τιμολόγιο είναι γύρω του, για την ενέργεια είναι 30% περίπου του εισοδήματος του νοικοκυριού και έχει γίνει ε, θέμα ακόμα πιο σημαντικό μετά την κρίση διότι το ποσοστό ε, της τιμολόγησης για την ενέργεια για κάθε οικογένεια έχει αυξηθεί και για την άμεση ενεργειακή αγορά και για τα αγαθά που αγοράζουμε στην, ε, στην αγορά. Υπάρχει εδώ μεγάλη ευκαιρία. Από ευρωπαϊκής απόψεως είναι, μιλάμε τώρα για 20% εξοικονόμηση το οποίο οδεύει προς αυτή την κατεύθυνση. Όταν βλέπετε ε, ποια είναι οι δύο τομείς για την εξοικονόμηση ενέργειας μπορούμε να πούμε ότι για αν ε, δείτε ότι είναι 100% η ενέργεια, 40% από τα 20% μπορούν να εξοικονομηθούν χρησιμοποιώντας τα έξυπνα ψηφιακά συστήματα για την εξοικονόμηση ενέργειας με ε, καλύτερη μετακίνηση στοιχεία, με καλύτερη κατανόηση στοιχείων μπορείτε κατά 40% ε, να βελτιώσετε από αυτό το 20%. Το άλλο 40% είναι στον τομέα της οικοδομής. Και στην οικοδομή τόσο το σύστημα θέρμανσης και η οικοδομή αυτή καθεαυτή είναι σημαντικά και νομίζω ότι είναι οι δύο ή τρει τομεί όπου μπορούμε να κάνουμε περισσότερο σε Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούμε με οδηγίες να αποφασίσουμε και να θέσουμε ορισμένα κριτήρια διότι πρέπει αυτό το 20% να επιτευχθεί μέχρι το 2020 αλλά αυτό δεν θα γίνει εκτός αν κάποιος εφαρμόσει αυτές τις αλλαγές και σε αυτούς τους τομείς οι εφαρμογές πρέπει να γίνουν από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και το μεγάλο θέμα που τίθεται τώρα έχουμε στον, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ολόκληρη την Ευρώπη τις δεξιότητες, τις ικανότητες για να γίνει αυτά. Αλλά υπάρχουν ε, χώρες, κυρίως από τα νέα κρατημέλη, όπως η δική μου χώρα, όπου οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν έχουν τέτοια μέσα, τέτοιες ικανότητες. Ε, υπάρχει αναλφιβητισμός ως προς τον χαμηλή κατανόλωση άνθρακα. Ο υδραυλικός, ο ηλεκτρολόγος δεν ξέρει να χρησιμοποιήσει την τεχνολογία που υπάρχει στην αγορά και ε, δεν ξέρει πώς να την χρησιμοποιήσει. Λέχθηκε επίσης σήμερα ότι η ενέργεια που δεν χρησιμοποιούμε είναι η φθηνότερη, αλλά είναι αληθές ότι είναι φθηνότερη. Όταν υπολογίσετε τις επενδύσεις που πρέπει να πραγματοποιηθούν και όταν πρέπει να γίνουν οι επενδύσεις, δεν μπορεί να είναι η φθηνότερη, τουλάχιστον για τα 10 πρώτα χρόνια όπου θα πρέπει να πληρωθεί η επένδυση και αυτό είναι ένα από τα μεγάλα κολλήματα και εμπόδια για να επιτύχουμε τον στόχο ενεργειακής απόδοσης. Πώς θα πείτε στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στα ευρωπαϊκά νοικοκυριά ότι αν τώρα επενδύσετε ορισμένα χρήματα σε 10 χρόνια θα αποδώσουν για σας. Και έχουμε αρκετά μέσα χρηματοοικονομικά για τέτοια έργα. Έχουμε ορισμένα κράτη-μέλη που μπορούν να το πράξουν, αλλά υπάρχουν ορισμένα κράτη-μέλη για τα οποία αυτές οι αντιλήψεις είναι σε υποανάπτυκτο στάδιο. Γι' αυτό οργανώνουμε εδώ στην Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τα Εθνικά Κοινοβούλια τέτοιες συναντήσεις για να μπορέσουμε να δώσουμε ευκαιρία ανταλλαγής απόψεων και νομίζω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να παίξει μείζωνα ρόλο προς την κατεύθυνση αυτή. Όταν μιλούμε για α, τις άλλη δυνητική εξοικονόμηση που είναι η έξυπνη τεχνολογία, έχουμε να αντιμετωπίσουμε άλλο πρόβλημα, διότι όταν μιλάμε για έξυπνη τεχνολογία το ότι υπάρχει σύγκρουση ανάμεσα στον παραδοσιακό ενεργειακό τομέα που, είναι, που έχει την τον βραδύτερο ρυθμό που την, έχει την βραδύτερη καμπύλη καινοτομία, ενώ όταν μιλάτε για τον τομέα των τεχνολογιών επικοινωνίας και πληροφορικής βλέπετε ότι, ε, ότι έχουμε τώρα τρίτης γενεάς κινητά τηλέφωνα ενώ το δίκτυο που έχετε στο σπίτι σας έχει τοποθετηθεί πριν από 20 χρόνια. Υπάρχει λοιπόν ανάμεσα στον παρδισιακό και στο σύγχρονο ε, κλάδο ε, σύγκρουση. Υπάρχουν διαφορετικές νομοθεσίες από το παρελθόν και αυτά τα πράγματα πρέπει να προσαρμοστούν. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα που θα είναι σημαντικό θέμα για το μέλλον. Αν έχετε έξυπνο σύστημα και αν έχετε ε, με το κινητό τηλέφωνο όλες τις πληροφορίες, όλα τα στοιχεία σας συλλέγονται και διοχετεύονται από το σύστημα. Ποιο σύστημα προστασίας δεδομένων πρέπει ε, να εισαγάγεται για να μην υπάρξει κακή χρήση, για να μπορεί ο καθένας ε, να δει αν ακολουθείτε την, το σωστό δρόμο και γιατί το κάνετε. Το, το σύστημα προστασίας δεδομένων ε, το τομέα ε, των τεχνολογιών επικοινωνίας και πληροφορικής θα είναι απαραίτητο και για τον ενεργειακό τομέα. Η ενεργειακή εξάρτηση δεν είναι μόνο για τους πόρους ε, που εξοικονομούμε είναι επίσης και οι, οικονομικές, οι οικονομικοί πόροι που διατίθενται για τον τομέα. Και εκεί έχουμε μεγάλο εμπόδιο στην Ευρώπη δεν έχουμε μόνο την εξοικονόμηση ενέργειας, χρειαζόμαστε χίλια δισεκατομμύρια επενδύσεων. Και παρόλο είχαμε το δεύτερο πακέτο, το τρίτο πακέτο νομοθεσία, το στόχο 20% για το 2020, 50% για το 2050 ή το πέρασμα στις εναλλακτικές πηγές για τα επόμενα χρόνια οι επενδύσεις σε μεγάλη κλίμακα δεν έχουν γίνει σε αυτόν τον τομέα και πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι ενώ δεν έχουμε τις επενδύσεις δεν μπορούμε να αλλάξουμε πολλά πράγματα διότι δεν θα αποδώσει η νομοθεσία, δεν θα αποδώσουν αυτά που έχουμε επί χάρτου, μόνο τα κατάλληλα έργα θα αποδώσουν και αυτό είναι σημαντικό για αυτούς που λαμβάνουν τις πολιτικές αποφάσεις εθνικά και ευρωπαϊκά να φτάσουμε στο σημείο που δεν θα μιλούμε μόνο, αλλά θα δράσουμε και ε, θα έχουμε αποτελέσματα. Γι' αυτό θα είναι σημαντικό. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό τελικά να πούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει αρμοδιότητα σχετικά με την ενέργεια. Η ενέργεια δεν είναι κοινοτική πολιτική από την συνθήκη της Λισαβόνας και γι' αυτό τα πράγματα είναι δύσκολα για ό,τι κάνουμε χρησιμοποιούμε άλλες κοινοτικές πολιτικές, στην περιβαλλοντική πολιτική, τα μέσα εσωτερικής αγοράς, την ε, πολιτική του ανταγωνισμού. Όταν προσπαθείτε να προσδιορίσετε το νερό ε, που είναι ενέργεια, το προσδιορίζετε με τη φιάλη, με το μπουκάλι με κάτι άλλο, όχι με την ίδια τη φύση του. Η ευθύνη των εθνικών κράτων που έχουν την αρμοδιότητα και την κυριαρχία απέναντι στην συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να κάνει κάτι. Η Ευρώπη δεν θα μπορέσει να επιτύχει το στόχο της ενώ τα εθνικά κοινοβούλια δεν καταβάλουν προσπάθειες για το σκοπό αυτό. Είμαι ευγνώμων που ήρθατε εδώ ε, χαίρομαι ε, που ήρθατε εδώ και ελπίζω να χαρείτε και τη μέρα σας στην Ευρώπη και στις ε, Βρυξέλλες και ελπίζω να βελτιωθεί η κατάσταση και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τα νοικοκυριά και όχι μόνο για τις μεγάλες βιομηχανίες. Szeretném Editet biztosítani, hogy én jól érzem magam itt, és nagyon örülök, hogy most hozzászólhatok ehhez a valóban stratégiai fontosságú témához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 Εν πάση περιπτώσει, εφόσον πρόκειται για ευφυή δίκτυα, θα πρέπει να σκεφτούμε και το πρόβλημα της ε, ε, συμπαραγωγής διότι στο κείμενο της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν γίνεται ικανά λόγος για αυτό το θέμα είναι κάτι όμως που υπάρχει στα μεγάλα αστικά δίκτυα η συμπαραγωγή και ε, πιστεύουμε ότι έχουμε, έχουμε και πρέπει να διατηρήσουμε αυτή την ιδιαιτερότητα, δηλαδή μεγάλα αστικά δίκτυα τα οποία χρησιμοποιούνται κυρίως για τη θέρμανση και κυρίως για το θερμό είδωρ μέσα στα κτίρια. Ε, εδώ τίθεται το τεράστιο πρόβλημα βέβαια της χρηματοδότησης, κάτι που αναφέρεται εξάλλου αρκετές φορές στο κείμενο. Αυτή η συμπαραγωγή είναι κάτι που μπορεί να μη θεωρηθεί παραγωγικό κάποια στιγμή εάν δεν υπάρχουν οι απαραίτητοι πόροι. Όμως μπορούμε να παράγουμε ταυτόχρονα θερμότητα και ηλεκτρικό ρεύμα. Και γι' αυτό θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας που του Δεν νομίζω ότι έχουμε το χρόνο να περατώσω ε, όλο μου το λόγο, να διαβάσω όλο μου το κείμενο. Ε, ε κύριε Φώτ, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, ευχαριστώ που μου δώσατε το λόγο στη σημερινή απογευματινή ε, συνεδρίαση. Το θέμα της ενέργειας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εγώ υπήρξα η εισηγήτρια εδώ στο Κοινοβούλιο ε, για τις διά... για τα, υπεράκτια δίκτυα και για τα όρια που παρουσιάζουν και αυτό ο στόχος της συζήτησης είναι να έχουμε φιέστερους τρόπους να διαχειριστούμε τη ζήτηση σε κοινοτικό επίπεδο. Η εξέταση της ζήτησης είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα σίγουρα, αλλά το όλο θέμα της ε, ασφάλειας εφοδιασμού, το θέμα της ποικιλομορφία και του ανταγωνισμού επίσης ε, κάτι το οποίο θα ενθαρρύνει την ασφάλεια του ε, εφοδιασμού αντιμετωπίζοντας και τις προκλήσεις. Όλα αυτά είναι σημαντικά τι θα κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, πού θα βρει τους πόρους, πώς θα βρει την χρηματοδότηση για, τα, για το αναξιοποιητό δυναμικό των δικτύων, ε, για την παροχή και, την, και τον εφοδιασμό της ενέργειας. Βλέπουμε ότι στην Ευρώπη όλο και πιο δυσχερές καθίσταται το να βρίσκονται πόροι για να χρηματοδοτούνται τα σχέδια που θέλουμε να εφαρμόσουμε. Τι θα κάνουμε λοιπόν, πώς θα διευκολύνουμε, ε, έχουμε εδώ ένα χάσμα ανάμεσα στα όνειρά μας και τους πόθους μας και την πραγματικότητα όταν θέλουμε να τα υλοποιήσουμε και ε, αυτές οι μακροπρόθεσμες επενδύσεις είναι επιθυμητές γιατί, γιατί ε, ε, υπάρχουν όσο περνάνε τα χρόνια ορισμένοι επενδυτές οι οποίοι αναζητούν τομείς για επενδύσεις. Εξετάζουμε λοιπόν όλους αυτούς τους τομείς, βλέπουμε όταν θέλουμε να δούμε πού θα βρούμε τα χρήματα για να ε, οικοδομήσουμε αυτό το σύστημα. Θα βάλουμε φραγμούς στο ίδιο μας το σύστημα για να, να φύγουν οι επενδυτές και να πάνε αλλού γιατί ε, θα πρέπει να δημιουργήσουμε μια ποικιλομορφία και να τους κρατήσουμε εδώ για τις ενεργειακές μας ανάγκες. Είναι αλήθεια ότι οι επενδυτές λένε ότι υπάρχει μια ανησυχία και η μεγαλύτερη ανησυχία τους είναι η αβεβαιότητα στο ρυθμιστικό πλαίσιο δεν ξέρουν ε, τι, πόσο μακροπρόθεσμο θα είναι στην πραγματικότητα αυτό το ενεργειακό σχέδιο. Τι θέλουμε λοιπόν, θέλουμε να καταρτήσουμε ένα πλαίσιο, να δουλέψουμε με, μαζί με διάφορες χώρες που έχουν ποικιλόμορφε ανάγκες και να είμαστε σίγουροι ότι έχουμε μία όσο πιο σταθερή βάση γίνεται. Ζούμε σε έναν αβεβαιό κόσμο, το παραδέχομαι, αλλά μπορούμε να φτιάξουμε μια σταθερή βάση όσο σταθερότερο γίνεται για να προσελκύσουμε κινητοποιήσουμε τους επενδυτές και του ιδιωτικού και του δημόσιου νέα για να συμμετάσχουν, να χρηματοδοτήσουν σε αυτή την, το σχέδια, αυτά τα σχέδια υποδομής μας. Εμείς θέλουμε να διασφαλίσουμε τον εφοδιασμό στην ενέργεια και να μην τη σπαταλούμε για το μέλλον. Αυτό είναι το μεγάλο μας όνειρο. Ευχαριστώ πολύ. Από την Αυστρία ο, ο Δόκτωρ Βίτμαν. Ε, εγώ επανέρχομαι επί του θέματος. Η, γιατί θέλω να σχολιάσω αυτά που είπε ο ε, συνάδελφος ε, Βίτμαν από την Πολωνία. Μας μίλησε για την εξοικονόμηση ενέργειας ε, στα συστήματα θέρμανσης που μας επιτρέπει μέχρι να φτάσουμε σε μια εξοικονόμηση της τάξης του 45 με 50% και έτσι να έχουμε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα σε ενεργειακό επίπεδο. Αυτό είναι ένα παράδειγμα που το είδαμε και στην Αυστρία. Εγώ θα ήθελα να έρθω στα, στις ορυκτές ε, πηγές ενέργειας. Ε, υπάρχει το πετρέλαιο επίσης, το φυσικό αέριο και όλα αυτά είναι περιορισμένα. Έχουμε προβλέψει πηγές ενέργειας οι οποίες δεν έχουν κανένα μέλλον σε 50 με 60 χρόνια. Δεν θα υπάρχει τίποτα από όλα αυτά, οπότε δεν κατανοώ γιατί πρέπει να επενδύουμε τεράστιους ε, πόρους ε, εφόσον δεν υπάρχει μέλλον. Είναι ευφυές αυτό. Ε, θα μειωθεί ε, μας υπόθηκε η κατανάλωση του φυσικού αερίου στα νοικοκυριά, υπάρχει ήδη μεγάλη πτώση και θα υπάρξει μεγαλύτερη χρήση των νέων τεχνολογιών. Οπότε ποια είναι η θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε σχέση με την μείωση του 30% μέχρι το 2020. Αν γίνει αυτή η μείωση θα έχουμε 14,2 Δύο δισεκατομμύρια ε, εξοικονόμηση και θα πρέπει να σταματήσει και αυτή η αλληλοεξάρτηση των δικτύων. Είμαστε εξαρτημένοι από τα ξένα δίκτυα, οπότε είναι αυτό ένα στοιχείο που πρέπει να το προσέξουμε ιδιαίτερως γιατί χρειαζόμαστε εισαγωγές. Εξαρτώμαστε από τις εισαγωγές πετρελαίου και δίνουν θέσεις εργασίας μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά εφόσον ε, καταργούμε θέσεις εργασίας σε χρειαζόμαστε ε, την, ε, τους εξωτερικούς συνεργάτες και χρειαζόμαστε συνεργασίες με τους έξω. Πρέπει να σας υπενθυμίσω ότι στο Φουκοσίμα έχουμε δυόμιση περίπου ε, φορές ε, ε, εκπομπές ρήπων περισσότερες από ό,τι είχαμε στο Τσέρνομπιλ. Κατανοείτε ότι αυτό είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα και ότι πρέπει να τα σκεφτούμε ε, όλα αυτά τα στοιχεία για να οικοδομήσουμε ένα πρόγραμμα ε, ε, σωστό πυρηνικό στην Ευρώπη μέσα στα επόμενα 20 με 30 χρόνια. Να έχουμε πολύ σωστές πυρηνικές εγκαταστάσεις είναι κάτι που αν θέλουμε να το πράξουμε μπορούμε, είναι απόλυτα εφικτό, θα είχαμε μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας. Ήδη το 20 με 30% του εφοδιασμού του ενεργειακού προέρχεται από, το πυρηνικό τομέα. Ε, θα μπορούσαμε να το προβλέψουμε με την Ευρατόμ αυτό το σχέδιο. Γιατί δεν έχουμε το δικαίωμα να το πράξουμε και ασχολούμαστε μόνο με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ε, το, η Ευρατόμ ε, απορρίπτεται από την κοινή γνώμη, έχει ένα 90% απόρριψη στην Αυστρία παραδείγματος χάρη. Ε, βλέπουμε όμως ότι υπάρχουν ανταγωνιστές στην παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος. Εμείς στην πατρίδα μου δεν μπορούμε να αγοράζουμε ηλεκτρικό ρεύμα από το εξωτερικό γιατί αποτελεί ένα τεράστιο οικονομικό πρόβλημα. Πρέπει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αντιδράσει σε όλα αυτά και πρέπει να έχουμε τη δυνατότητα σε όλα τα στρώματα του πληθυσμού να ε, παρέχουμε ε, ένα σωστό εφοδιασμό ε, ενέργειας. Επίσης υπάρχει το ενεργειακό μείγμα της Ένωσης. Σε αυτό θέλω να αναφερθώ. Πολύ συχνά υπόθηκε ότι είναι εθνική υπόθεση. Εάν υπάρχουν ακτινοβολίες όμως δεν είναι εθνικό θέμα. Εάν είναι επικίνδυνες οι ακτινοβολίες ε, πρέπει να αλλάξει το ενεργειακό μίσμα της Ένωσης γιατί πρόκειται για το μέλλον μας. Ευχαριστώ πολύ για την ε, παρέμβασή σας. Τώρα θα μιλήσουμε για τα ευθυνή e συστήματα. Δεν πρόκειται εδώ να μιλήσουμε πολύ για την ε, πυρηνική ενέργεια, διότι διότι τώρα θα ήθελα να δώσω τον λόγο στον κύριο Γιάνκου από την ε, Ρουμανία. Ευχαριστώ πολύ. Κατά τη γνώμη μου, το θέμα αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό και θα ήθελα να τονίσω μερικές απόψεις που δεν αναφέρθηκαν μέχρι τώρα. Θα ήθελα να μιλήσω για το γεγονός ότι η ενέργεια προϋποθέτει μια ανάλυση των ενεργειακών δικτύων ως ζώντα δίκτυα. Για να έχουμε ζώντα δίκτυα θα πρέπει να έχουμε υψηλό επίπεδο επενδύσεων σε νέες τεχνολογίες και εδώ έχουμε να αντιμετωπίσουμε δύο προκλήσεις. Πρώτα απ' όλα μια αύξηση της κατανάλωσης ενέργειας. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Διεθνούς Υπηρεσίας Ενέργειας, η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας θα διπλασιαστεί κατά 18.000 τεραβάτ θα περάσει σε 34.000 τεραβάτ ανά ώρα. Αυτό προϋποθέτει προσπάθεια ε, επενδύσεων 21 τρισεκατομμυρίων δολαρίων. Η ίδια η Ευρώπη ανέπρεπε να αυξήσει την ενεργειακή της κατανάλωση και να τροφοδοτήσει, να εφοδιάσει αυτή την ε, ε, πρόσθετη κατανάλωση με ενεργειακούς πόρους θα χρειαζόταν ε, έναν δρόμο από τις Βρυξέλλες μέχρι το Πεκίνο ε, με εγκαταστάσεις αιωλικής ενέργειας από τις δύο πλευρές και εκατομμύρια ε, ποδοσφαιρικών γηπέδων που να καλύπτονται από ε, φωτοβολταϊκά συστήματα. Χρειαζόμαστε λοιπόν υλικό, εξοπλισμό που να πηγαίνει μέχρι τον καταναλωτή και που να επιτρέπει στον καταναλωτή να ελέγξει την κατανάλωση ενέργειας. Πρώτη πρόκληση είναι η ανθρώπινος πόρος η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει να αντιμετωπίσει ένα μείζον πρόβλημα. Είναι η γύρανση του πληθυσμού και δεύτερον η νέα γενεά δεν έχει κλείσει τάση να μελετάει τεχνικά προφίλ. Νομίζω ότι σε όλα τα κράτη-μέλη έχουμε ε, έλλειψη επαγγελματιών και εμπειρογνωμοσύνη στον ενεργειακό τομέα, διότι χρειάζονται ειδικέ γνώσεις, ειδικοί εμπειρογνώμονε, ακόμη περισσότερο για τα ευφύ δίκτυα. Έχουμε πρόβλημα. Οι ανθρώπινοι πόροι είναι τρωτοί, ευάλωτοι. Έχουμε επίσης συμφόρηση στην παραγωγή τεχνολογίας θα πρέπει κάθε χρόνο να αντικαθιστούμε 25% της δυναμικότητας που υπάρχει, να ανακαινίζουμε τα δίκτυα μεταφοράς, να έχουμε νέες τεχνολογίες και αυτόματα συστήματα. Μια, ένα τρίτο τροτό σημείο είναι ο πόρος, ο χρηματοοικονομικός. Δύο παραδείγματα δόθηκαν και θα ήθελα να τα τονίσω. Πρόκειται για την θερμική ενέργεια. Ο τομέας αυτός εγκαταλείφθηκε τα 20 τελευταία χρόνια στο επίπεδο των κρατών μιλών, κυρίως από τα κράτη-μέλη ε, του κέντρου και της νότιο-ανατολικής Ευρώπης και χάσαμε την τοπική αγορά θερμικής ενέργειας. Ο πληθυσμός αναγκάστηκε να αποσυνδεθεί ε, διότι οι τιμές ήταν πάρα πολύ ψηλές. Ε, Όλα αυτά προϋποθέτουν σύμφωνα με την γνώμη των ειδικών του ενεργειακού τομέα ε, είχα μιλήσει πριν για μια μελέτη της Διεθνούς Υπηρεσίας Ενέργειας. Η πρώτη προτεραιότητα των ειδικών είναι η ενεργική, ενεργειακή απόδοση, μια μελέτη που έχει γίνει σε 84 κράτη σε ολόκληρο τον κόσμο. Η απόδοση, η αποδοτικότητα ενεργειακή πρέπει να είναι η πρώτη προτεραιότητα των επενδυτών σε παγκόσμιο επίπεδο. Σε χώρες όπως η Ρουμανία, οι δυνατότητες μείωση κατανάλωσης είναι κατά 50%. Η Ρουμανία ε, καταναλώνει 40% της ενέργειας στα κτίρια και η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας αντιπροσωπεύει 70% του προϋπολογισμού ενός νοικοκυριού κυρίως το χειμώνα. Κατά τη γνώμη μου είναι υποχρεωτικό να ε, σχεδιάσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο ε, χρηματοοικονομικά συστήματα για την μεταφορά προχωρημένης τεχνολογίας, για συμπαραγωγή ε, και μεταφορά από την βόρειο-δυτική Ευρώπη προς την νότιο-ανατολική Ευρώπη, διότι το κέντρο και η νότιο-ανατολική Ευρώπη χρειάζονται υψηλή αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα στην χρησιμοποίηση της ενεργειακής ύλης. Πρέπει να έχουμε μια ενιαία, μια μοναδική θεώρηση από τα κράτη-μέλη, διότι είναι τα κράτη-μέλη που εξασφαλίζουν ε, την ανάπτυξη και την ισορροπία του ενεργειακού ε, ισολογισμού. Χρειαζόμαστε εθνικό παρατηρητήριο που να έχει εκπροσώπους σε εθνικό επίπεδο. Χρειαζόμαστε παρακολούθηση όλων των κοινοβουλίων για να θέσουμε τις βάσεις των απαιτουμένων στρατηγικών σχεδίων. Και τρίτον, πρέπει να προσδιορίσουμε τους χρηματικούς μηχανισμούς για την μεταφορά τεχνολογίας ανάμεσα στα κράτη-μέλη και επίσης για να αξιοποιήσουμε την αγορά εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Και τώρα ε, θα δώσω τον λόγο στον κύριο Παρακόσκας από την Λιθουανία. Ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί ε, συνάδελφοι, θα ήθελα να αντιδράσω σε αυτά που είπε ο κ. Βίτμαν από την Αυστρία. Και αντιδρώντας θα ήθελα ε, πρώτα απ' όλα να τονίσω την ιδέα ότι όταν μιλάμε για ενεργειακή ασφάλεια, για πυρηνική ασφάλεια μάλλον, δεν θα πρέπει να μιλούμε μόνον ε, για την διαχείριση των πυρηνικών σταθμών και μονάδων, αλλά επίσης και για τους ε, πυρηνικούς σταθμούς που κατασκευάζονται πολύ κοντά στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ρωσία και η Λευκορωσία προγραμματίζουν να κατασκευάσουν δύο πυρηνικές μονάδες που δεν θα είναι μακριά από την Λιθουανία που είναι σύνορο της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά την τραγωδία της Φουκοσίμα έχουμε συνειδητοποιήσει ότι η πυρηνική ενέργεια δεν είναι εξίσου ασφαλής όσο μας είπαν τις δύο τελευταίες δεκαετίες. Σε περίπτωση ατυχήματος στο μέλλον η πυρηνική σταθμή στην Ρωσία και στην Λευκορωσία ε, σε τέτοια περίπτωση η ρήπανση θα έφτανε στην Βαλτική θάλασσα διαμέσου των ποταμών της Λιθουανίας και θα έφτανε στη Δανία, στην Σουηδία ε, και σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Συνεπώς, νομίζω ότι οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι αντίστοιχα όργανα θα πρέπει να είναι προδραστικά σε αυτές τις περιστάσεις, διότι η Λιθουανία μόνη της δεν θα μπορέσει να αντιμετωπίσει αυτά τα θέματα ενεργειακής ασφάλειας. Ούτε θα μπορεί μόνη της να εξασφαλίσει ε, την ασφάλεια ολόκληρης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί μιλούμε γι' αυτό, γιατί η κατάσταση ούτε στη Ρωσία ούτε στην Λευκορωσία δεν είναι ρόδινη από αυτή την άποψη. Ευχαριστώ. Τώρα δίνω τον λόγο στο συνάδελφο Οντί. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η παρέμβασή μου σχετίζεται με τις υποδομές σχετικά με τον εφοδιασμό τον ενεργειακό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται σε Ήπειρο και Είμαστε σε ανταγωνισμό με άλλες υπήρους, αλλά με μία διαφορά είναι ότι οι ανταγωνιστές μας είναι κράτη και εμείς είμαστε μια ένωση κρατών. Έχουμε να ανταγωνιστούμε την Κίνα, τη Βραζιλία, την Ινδία, τη Ρωσία, τις Ηνωμένε Πολιτείε που είναι κράτη. Εμείς είμαστε μια ένωση κρατών, θα πρέπει πρώτα να συμφωνήσουμε μεταξύ μας προτού η πραγματικότητα να γίνει ευρωπαϊκή και ως προς τις υποδομές τις ενεργειακές, οι οποίες είναι ένα στοιχείο ανταγωνιστικότητας του Ισυπήρου μας, θα ήθελα να προτείνω την ιδέα της διαχείρισής τους και του μέλλοντός τους διότι αφότου απελευθερώσαμε την αγορά ενέργειας δεν ξέρουμε πολύ καλά πού είναι τα δίκτυα και ποιοι είναι οι διοκτήτες των δικτύων. Είχαμε κύριε Πρόεδρε ε, μία συνεδρίαση για τις απαιτούμενε επενδύσεις στις ενεργειακές υποδομές και έθεσα την ερώτηση, υπήρχαν εκεί πολλοί ειδικοί ειδικοί ιδιοκτήτε αερίου, η Gaz de France και ρώτησα ποιος είναι ο ιδιοκτήτη των δικτύων. Κανείς σήμερα δεν ξέρει ποιος είναι ο ιδιοκτήτη των δικτύων. Και αν κάποιο, η Gazprom, αρχίζει να αγοράζει δίκτυα με ενό άλλου κράτου, ποιο θα εμποδίσει την Gazprom. Ήθελα να επισύρω την προσοχή σα πάνω στο θέμα αυτό, διότι οι συμπολίτε μα δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Του εκπροσωπούμε, εκπροσωπούμε του Ευρωπαίου πολίτε και νομίζω ότι έχουμε καθήκον να εξασφαλίσουμε την ποιότητα των δικτύων, την ασφάλεια των δικτύων, την διασύνδεση ανάμεσα στα κράτη-μέλη, την ανεξαρτησία, την πολιτική της ιδιοκτησίας των δικτύων και αυτό και αυτήν την ασφάλεια πρέπει να την μεταδώσουμε και την διαβεβαίωση αυτή στους συμπολίτες μας. Διαρωτώ με μήπως ήρθε η στιγμή να διαπραγματευτούμε με τους φορείς, με τους οργανισμούς, ούτως ώστε το σύνολο των ευρωπαϊκών δικτύων να ανήκει σε μια μεγάλη ευρωπαϊκή εταιρεία ενεργειακών δικτύων που θα είχε ως αποστολή να διατηρήσει τις διασυνδέσεις, να κάνει τις επενδύσεις βεβαίως με τις αρχές τιμολόγησης, ε, να επιβαρύνει την κατανάλωση με το κόστος και να υπάρξει κάποια αλληλεγγύη αλλά να δώσει στην Ήπειρο την ασφάλεια ότι έχουμε την καλύτερη παραγωγικότητα, την καλύτερη εξυπηρώτηση, ότι ο κάθε καταναλωτής Ευρωπαίος θα εξυπηρετείται όπου και αν βρίσκεται στο ευρωπαϊκό έδαφος, τόσο ώστε να έχουμε τον καλύτερο λόγο ε, τιμής ποιότητας με την αποτελεσματικότητα την οικονομική, με ε, μηχανικούς ε, υψηλού ε, επίπεδου διεθνούς για να εξασφαλίσουμε την Ήπειρό μας βεβαίως. Οι οργανισμοί μετά θα ανταγωνίζονται για την παραγωγή και την διανομή ενέργειας. Αυτή είναι η ιδέα που καταθέτω. So, danke sehr. Ich habe jetzt äh, eine letzte Wortmeldung. Äh, oh. Ah. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κατά τη διάρκεια όλων αυτών των συζητήσεων Νομίζω ότι δύο είναι τα μεγάλα θέματα που προέκυψαν. Ε, το πρώτο θέμα είναι ο ανεφοδιασμός, ο εφοδιασμός στην ενέργεια και ε, δεύτερον η κατοχύρωση της ασφάλειας ε, ε, του εφοδιασμού ειδικά στον πυρηνικό τομέα. Δηλαδή ότι πρέπει να λάβουμε υπόψη τον πυρηνικό τομέα πάρα πολύ σοβαρά. Ένα τρίτο στοιχείο που θα ήθελα εγώ να θίξω είναι οι νέες τεχνολογίες και οι νέες έρευνες. Ακούστηκε ήδη ότι μπορούμε να εξοικονομήσουμε πάρα πολύ ενέργεια εάν ε, χρησιμοποιήσουμε την γεωθερμική μέθοδο. Υπάρχουν έρευνες ε, την παρούσα στιγμή. Πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να εξοικονομήσουμε με τον καλύτερο τρόπο την περισσότερη ενέργεια. Πάρα πολύ συχνά βλέπουμε ότι οι εξοικονομήσεις αυτές είναι αποτελεσματικές. Βλέπουμε τις ηλεκτρικές συσκευές ε, παραδείγματος χάρη ότι πρέπει να, να βγάζουμε την πρίζα ή να, να, ε, ε, να σβήνουμε ε, εντελώς τις συσκευές και έτσι κάνουμε μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας ενώ αφήνουμε συνήθως το stand-by τη συσκευή και δεν σβήνουμε το διακόπτη έτσι χάνεται πάρα πολύ ενέργεια αυτό είναι ένα μικρό παράδειγμα που μας δείχνει ότι πόσο πρέπει να είμαστε ενημερωμένοι σε όλους αυτούς τους τομείς και πώς θα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις εξοικονομικές την εξοικονόμηση ενέργειας που θα κάνουμε νέες πηγές ενέργειας. Ευχαριστώ πολύ. Ε, η κυρία Βερσισόρ έχει το λόγο ως εισηγήτρια. Ε, ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ανακεφαλαιώσω ορισμένα σημεία πριν από το πέρας της σημερινής συζήτησης, τουλάχιστον για να μπορέσουμε να έχουμε τις σωστές διαπραγματεύσεις στη συνέχεια. Ο τελευταίος ομιλητής παρατήρησα ότι είπε ε, για ένα, ότι υπάρχει ένα κενό στην έρευνα και στην ανάπτυξη. Γι' αυτό αποφασίσαμε να ε, ακολουθήσουμε ένα σχέδιο, μια νέα στρατηγική ε, ανάπτυξης ε, και ενέργειας αλλά χρειάζεται χρηματοδότηση. Χρόνια πριν είχαμε αποφασίσει να δράσουμε κατά αυτόν τον τρόπο. Υπήρχε ο κύριος Χατζόκ ήταν σκιώδης εισηγητής ε, στην ε, σχετική εισήγηση που είχε αναλυθεί από την Σοσιαλιστική Ομάδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και υπήρχαν προβλήματα χρηματοδότησης. Ε, το κόστος των 18 δισεκατομμυρίων για το σχέδιο έρευνας ε, βλέπετε ότι δεν μπορεί να αποδοθεί, δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί. Πρέπει να βρούμε έναν καλύτερο τρόπο, πρέπει να ε, υπάρξει χρηματοδότηση του σχεδίου τεχνολογίας για να μπορέσουμε να περάσουμε από την έρευνα στην εφαρμογή. Χρειάζεται ένας κοινό στόχος. Ο στόχος μας είναι να καταργήσουμε ε, ε, ρυθμιστικά τους φραγμούς. Αυτό δεν είναι μόνο ένα εθνικό πρόβλημα, ούτε ένα περιφερειακό. Υπάρχει και το επίπεδο της τοπικής αυτοδιοίκησης που είναι πάρα πολύ σημαντικό και εκεί υπάρχουν μεγάλοι φραγμοί. Ε, ο κύριος Γιουζάν άφερε ε, το κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι ε, το κείμενο των συναλλαγών προέκυψε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο για να μπορέσει να υπάρξει μια σωστή χρηματοδότηση όλων αυτών των σχεδίων για να υπάρξουν στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό περισσότερες παροχές ούτως ώστε να μπορεί να εφαρμόσει περισσότερα τέτοια σχέδια. Όλες οι χώρες μέλη ασκούν επικρίσεις, είναι πάρα πολύ κριτικές στο θέμα της χρηματοδότησης, δεν κατανοούν όμως ε, το πώς πρέπει να δράσουμε. Τι θα κάνουμε για την εξοικονόμηση ενέργειας, είναι έργο του Υπουργείου Οικονομικών αυτό, τι θα, το, θα αναλάβουν τις πρωτοβουλίες οι Υπουργοί Οικονομικών. Δεν νομίζω. Νομίζω ότι εμείς πρέπει να τις αναλάβουμε. Ένα άλλο σημείο που είναι πολύ σημαντικό είναι τα ευφύ δίκτυα και πιστεύουμε ότι στο κοινοβούλιο μας θα γίνουν ε, πολύ σωστές, θα ληφθούν σωστές αποφάσεις για εξοικονομήσεις και ε, πρέπει τα μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί για το είδωρ και για το ηλεκτρικό ρεύμα θα πρέπει να μεταφερθούν από τον τομέα των οικοκυριών που είναι ένας σκοτεινός τομέας ε, σε έναν τομέα ε, με ψηφιακούς δείκτες, με ένα κεντρικό σύστημα για να βλέπουμε αμέσως τις εξοικονομήσεις που γίνονται, για να βλέπουμε αμέσως πόσες ε, ε, εξοικονομήσεις κάνουμε. Ο περισσότερος κόσμος δεν ενδιαφέρεται για αυτά τα πράγματα. Όταν όμως δει ότι εξοικονομούμε ένα ευρώ την ώρα με ορισμένα συστήματα θα καταλάβει ότι μέσα στα επόμενα δέκα χρόνια η διαφορά θα είναι τέτοια η οποία θα γίνεται με βάση τις εξοικονομήσεις των οικοκυριών που θα ωφελήσει την Ευρώπη ολόκληρη. Α, θα περατώσω σε αυτό το σημείο επαναλαμβάνοντας αυτά που είπα και στην αρχή. Ήταν η πρώτη φορά που είχαμε μια τέτοια συζήτηση, πάρα πολύ θετική. Πρέπει να συνεχίσουμε για να δούμε σε νομοθετικό επίπεδο τι θα γίνει. Αν ο Ευρωπαίος νομοθέτης μαζί με τον Εθνικό νομοθέτη θα μπορέσουν να βρουν έναν σύνδεσμο τους ώστε να διαβιώσουν σε καμιά, να ζήσουν μια καλύτερη ζωή οι πολίτες μας. Το λόγο τώρα έχει ο κύριος Κόβατ. Θα έχει τον τελευταίο λόγο για αυτό το ζήτημα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, ευχαριστώ πολύ που μου δώσατε το λόγο. Το μικρόφωνο σας παρακαλώ το μικρόφωνο. Ένα λεπτό υπάρχει ένα τεχνικό πρόβλημα. Έλεγα λοιπόν, λέει ο κύριος Κόβατς, ότι επρόκειτο να μιλήσω στην μητρική μου γλώσσα για να ε, περατώσω αυτή την πάρα πολύ ενδιαφέρουσα απογευματινή μας συζήτηση θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι σε επίπεδο πολιτικών αποφάσεων αλλά και σε τεχνικό επίπεδο ε, οι ίδιες συζητήσεις πάντα γίνονται ε, και στη χώρα μας και πραγματικά όλα τα θέματα τα οποία εφήγησαν κατά τη διάρκεια αυτής της συζήτησης θα τα συζητήσουμε, θα τα διαβιβάσουμε στον αρμόδιο Υπουργό ούτως ώστε να μπορέσουν να συζητηθούν ε, όλα αυτά τα θέματα και σε εθνικό επίπεδο. Ε, υπήρξαν ορισμένα ενδιαφέροντα ερωτήματα. Ένα από αυτά ήταν αν χρειάζονται ευρωπαϊκές υποδομές όπως προβλέπεται και εδώ πρέπει να πω ότι η Προεδρία θεωρεί ότι το πρόβλημα δεν είναι καθόλου ότι έχουμε μη απαραίτητε δομές ή ότι έχουμε ε, λάβει περιτά μέτρα για, ε, την, ε, για τον εφοδιασμό μας. Γιατί δεν έχουμε τεράστια αποθέματα. Τα αποθέματα θα πρέπει να μπορούν ε, να κυκλοφορούν από τη μία περιφέρεια της άλλης στην Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί έτσι μειώνεται και το πρόβλημα της εξάρτησης. Ε, οπότε πρέπει να αναπτυχθούν οι υποδομές για να μπορούμε να έχουμε αποθέματα από κοινού δυνάμει. Και αυτό είναι κάτι το απαραίτητο. Για να αναπτύξουμε λοιπόν αυτές τις υποδομές προβλέπουμε μια πρώτη φάση χρηματοδότησης από την αγορά. Στην πρώτη φάση λοιπόν χρηματοδοτεί η αγορά. Ή μάλλον αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι δεν θα είναι μόνο η χρηματοδότηση της αγοράς αλλά θα υπάρχει και μια παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ταυτοχρόνως ούτως ώστε να δείξουμε πόσο αποτελεί προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση το θέμα αυτό. Πιστεύουμε ότι θα μπορούσαμε όλοι μας να συμφωνήσουμε στο ότι η πιο οικονομική ενέργεια, η πιο φτηνή τέλο πάντων, είναι η ενέργεια την οποία δεν καταναλώνουμε. Παρ' όλα αυτά πρέπει να διασφαλίσουμε να κατοχυρώσουμε την ασφάλεια του εφοδιασμού, να έχουμε δίκτυα τα οποία λειτουργούν και μία αποτελεσματικότητα των δικτύων η οποία μπορεί να βελτιωθεί εάν οι χρήστες ή τουλάχιστον οι τελικοί χρήστες είναι σίγουροι ότι μπορούν να υποφεληθούν ε, στην κατανάλωση. Επίσης πρέπει να παράγουμε ενέργεια, ένα μικρό μέρος της ενέργειας και τα πλεονάσματα που δεν θα χρησιμοποιηθούν θα μπορούν να επιστρέφονται στο δίκτυο. Ε, επίσης υπάρχουν οι ευφυείς μετρητές. Αυτό είναι ένα ενδιάμεσο σύστημα πάρα πολύ σημαντικό. Όλα τα ευφυείς συστήματα πρέπει να αναπτυχθούν περαιτέρω και μέσα στο πλαίσιο των ευφυών δικτύων ε, και της εφαρμογής τους είδαμε κάτι πολύ σημαντικό. Είδαμε ένα σημαντικό σημείο ότι χρειάζεται διαδραστικότητα, ότι πρέπει να ενθαρρύνουμε την διαδραστικότητα μεταξύ των επιχειρήσεων που ε, εφοδιάζουν και τους καταναλωτές. Μόνον έτσι θα γίνει δυνατό να υπάρχει πλήρης ολοκλήρωση και των ανανεώσιμων ε, ε, πηγών ενέργειας στο νέο σύστημα. Ένα άλλο σημαντικό σημείο το οποίο δεν ακούστηκε σήμερα το απόγευμα τουλάχιστον άμεσα ε, είναι το εξής. Πρέπει να δούμε σε ποια στιγμή θα υπάρξει γενίκευση των ηλεκτρικών οχημάτων γιατί αυτό θα έχει σίγουρα επίπτωση στην κατανάλωση βεβαίως και στις ανάγκες ηλεκτρικού ρεύματος οι ενεργειακές αγορές είναι πολύ στενά συνδεδεμένες μεταξύ τους και η απόφαση που λαμβάνει ένα κράτος είναι πάρα πολύ σημαντική, έχει επιπτώσεις άμεσες ε, στα γειτονικά κράτη και βεβαίως επηρεάζει τους, τη ζωή των καταναλωτών. Πέρα από αυτό μπορούμε να πούμε δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ το θέμα της ανταγωνιστικότητας και τον αντίκτυπο που έχουν όλα αυτά στην ίδια την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης όχι μόνο για το θέμα ε, της παραγωγής πυρηνικής ενέργειας για παράδειγμα αλλά και για το θέμα των πυρηνικών αποβλήτων πολλές ευρωπαϊκές εταιρείες απορρίπτουν αυτή την επιλογή, απορρίπτουν καθαρά την πυρηνική ενέργεια. Εμείς πιστεύουμε ότι πριν να λάβουμε την οποιαδήποτε απόφαση πρέπει να οργανώσουμε μια πολύ ευρεία συζήτηση για να δούμε ε, την συνένεση την ενδεχόμενη. Είναι ο μόνος τρόπος να συμβάλλουμε σε μια μεικτή ανάπτυξη όλων των πηγών ενέργειας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Κόβατς για την παρέμβασή σας και Ευχαριστώ όλους τους αγορητές αλλά και όλους τους παρόντες για τις πολύ χρήσιμες ε, και αποδοτικές συμβολές σας που ακούσαμε αυτές τις τρεις τελευταίες ώρες. Περατώνοντας θα ήθελα να σας πω και την γνώμη μου, την άποψή μου. Θεωρώ ότι υπάρχει μια κοινή στάση, μια κοινή θέση για, σε σχέση με όλα όσα ακούστηκαν σήμερα. Ένα είναι το μεγάλο θέμα, η διασύνδεση. Ε, υπάρχουν πολλά επιχειρήματα υπέρ της διασύνδεσης γιατί ε, έτσι έχουμε λιγότερη εξάρτηση σε ενεργειακό επίπεδο. Είναι κάτι το απαραίτητο το να είμαστε συνδεδεμένοι ε, να είναι συνδεδεμένα τα δίκτυα τα ευρωπαϊκά ε, και γιατί έχουμε πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο ως Ευρώπη δηλαδή σε σχέση με ε, τους έξω. Γι' αυτό νομίζω ότι τα δίκτυά μας πρέπει να έχουν διασυνδέσεις. Δεν έχουμε εναλλακτικέ ενεργειακές οδούς. Και θα έλεγα λοιπόν ότι σήμερα Συμφωνούμε όλοι μας στο ότι πρέπει να επιτύχουμε αυτόν τον στόχο της διασύνδεσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο και επίσης χρειαζόμαστε ευρωπαϊκούς πόρους χρηματοδότησης. Πέρα από αυτό ακούσαμε πάρα πολλά καλά και σωστά επιχειρήματα στην απογευματινή μας συνεδρίαση και Ίσως θα πρέπει να μπορούμε κάποια στιγμή να γίνουμε πλήρως ανεξάρτητοι από την ενέργεια που προέρχεται από τρίτες χώρες. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μπροστά της ένα μακρύ δρόμο ε, αλλά νομίζω ότι μπορούμε τουλάχιστον σε μια πρώτη φάση να περιορίσουμε τα μέγιστα αυτήν την εξάρτηση και να δράσουμε κάνοντας μερικά θετικά βήματα, βρίσκοντας εναλλακτικές λύσεις. Επίσης, η κατανομή των ε, αρμοδιοτήτων μεταξύ Ευρώπης και κρατών μελών είναι ένα καινούριο θέμα, το οποίο κανονικά δεν έπρεπε να το θίξουμε σήμερα. Ορισμένοι όμως το έθιξαν, το θέμα των Εθνικών Κοινοβουλίων και των σχέσεών τους με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έχουμε έναν ελάχιστο στόχο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αυτό είναι σαφές σε σχέση με τις ε, πηγές των, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ε, σε σχέση με το ενεργειακό μείγμα της Ένωσης και το ενεργειακό μείγμα των κρατών μελών. Η Ένωση λοιπόν έχει και πρέπει και μπορεί να διαδραματίσει ένα ρόλο. Ε, ίσως να είμαστε να πρέπει να είμαστε περισσότερο σύμφωνοι σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Νομίζω ότι το Φοκουσίμα ε, παίζει ένα ρόλο πάρα πολύ σημαντικό στο να συνενέσουμε και υπάρχουν και άλλα θέματα που ακούστηκαν οι δύο ενέργειες παραδείγματος χάρη, ε, οι εναλλακτικές πηγές για η Επιτροπή Αποβλήτων για ορισμένα κράτη-μέλη, το θέμα της ε, κατανάλωσης ε, των υδρογονανθράκων που δημιουργεί προβλήματα σε ορισμένες άλλες περιφέρειες και όπως λέγαμε θέμα της καύσης των αποβλήτων τέθηκε, πολύ σημαντικό θέμα και τα λοιπά. Κατά αυτόν τον τρόπο βλέπουμε ότι υπάρχουν θέματα που προκαλούν αντιθέσεις και αντιφάσεις κατά τη διάρκεια των συζητήσεων. Ίσως ε, υπάρχει και κάτι το οποίο δεν το θίξαμε, δεν μιλήσαμε καθόλου γι' αυτό. Είναι το θέμα της εξέλιξης των ευρωπαϊκών δικτύων. Είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά τα δίκτυα για το μέλλον της Ευρώπης, πάρα πολύ. Και γι' αυτό θα ήθελα να υπογραμμίσω την, ε, συμφο... την σημασία των εφιών δικτύων και ξέρουμε ότι σε πάρα πολλές χώρες ε, καταφεύγουμε σε μια μέση κατανάλωση για να γίνεται μια αξιολόγηση θεωρητική της κατανάλωσης, ένας υπολογισμός ε, που δεν επιτρέπει την εξοικονόμηση της ενέργειας για να δεν, δεν μας επιτρέπει να λάβουμε πρωτοβουλίες μέσα στα νοικοκυριά για να μειώσουμε την ε, κατανάλωση της ενέργειας όταν πληρώνουμε βάσει ενός γενικού υπολογισμού. Οπότε πιστεύω ότι αυτοί οι στόχοι πρέπει να ξεκαθαριστούν γιατί έχουν μεγάλη σημασία. Ένας στόχος ε, που δεν είναι μόνο εθνικός αλλά είναι και ευρωπαϊκός μας αφορά όλους. Το θέμα το υπογράμμισαν πάρα πολλοί αγορητές και ελπίζω ότι μπορούμε να περατώσουμε λέγοντας ότι η επόμενη επόμενες προεδρίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, θα ξαναδούν αυτά τα θέματα μέσα στα πλαίσια των εργασιών τους. Αυτά ήθελα να σας πω αγαπητοί συνάδελφοι. Τα συμπεράσματά μου ίσως είναι λίγο υποκειμενικά σε σχέση με τη σημερινή μας συζήτηση. Θα ήθελα να ξαναδώσω τώρα τον λόγο στον κύριο Γκιούρκ που ίσως έχει μερικές παρατηρήσεις να υποβάλει. Θα προσπαθήσω να συνοψίσω τις ε, συζητήσεις των τριών τελευταίων ώρων. Θα είναι δύσκολο βέβαια πώς να συνοψίσει κανείς τρεις ώρες συζήτησης μέσα σε λίγα λεπτά. Ε, ε, βεβαίως ε, δεν θέλω να μακρηγορήσω, θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος αλλά να κάνω μια πλήρη σύνοψη των συζητήσεων. Αρχίζοντας θα ήθελα να ευχαριστήσω τους βουλευτές των Εθνικών Κοινοβουλίων που έκαναν την προσπάθεια να έρθουν μέχρι εδώ για να συμμετάσχουν στη σημερινή συζήτηση. Η συζήτηση αυτή είναι πάρα πολύ σημαντική για μας στο Κοινοβούλιο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους εσάς που μείνατε μέχρι το τέλος της συζήτησης και πιστεύω ότι η απόφαση του Κοινοβουλίου και το, του Εθνικού Κοινοβουλίου της Ουγγαρίας για τη διοργάνωση της σημερινής μεικτής συνεδρίασης ήταν μια πάρα πολύ καλή ιδέα δεδομένη της κρίσης ε, οικονομικής και χρηματοπιστωτικής που βιώνουμε βεβαίως. Μπορούμε να συζητήσουμε για πάρα πολλά ζητήματα, αλλά ήδη το ενεργειακό ζήτημα είναι κέριο. Η Ουγγρική Προεδρία ούτως ή άλλως έχει αναδείξει αυτό το θέμα σε προτεραιότητα, το αναφέραμε πολλές φορές κατά τη διάρκεια της συζήτησης και γι' αυτό το λόγο επιλέξαμε το σημερινό θέμα για την μεικτή συνεδρίαση. Πρόσφατα συγκαλέσαμε ένα, ε, μια συνεδρίαση ε, στο Συμβούλιο αποκλειστικά και μόνο για ενεργειακά ζητήματα. Ε, πρώτη φορά γινόταν αυτό, το 2004. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, α και να πω ότι τότε εξελέγει βουλευτής, Τότε λοιπόν η Επιτροπή Βιομηχανίας δεν είχε πάνω στα φώτα της δημοσιότητας, δεν ήταν αν θέλετε ε, δημοφιλής ε, επιτροπή εκείνη την εποχή. Όμως με την ε, κοινή ενεργειακή πολιτική που σταδιακά εκπονήθηκε τα τελευταία χρόνια άλλαξε η κατάσταση. Η ενεργειακή ασφάλεια, η σταθερότητα στον εφοδιασμό και οι λογικές τιμές ε, τελικά είναι τα βασικότερα ζητήματα. Τότε επίσης δεν ήταν και ιδιαίτερα ελκυστικό αν θέλετε το ζήτημα. Όμως ε, οι πρόσφατες ε, εξελίξεις, παραδείγματος χάρη μεγάλες διακοιμάσεις τιμής του πετρελαίου, η κατάρρευση των χρηματοπιστωτικών αγορών και άλλες τέτοιες εξελίξεις τροποποίησαν τα δεδομένα και αντιλαμβανόμαστε πως ε, προέκυψαν ε, προσφορότατες ε, προτάσεις από τον ίδιο τον ενεργειακό κλάδο για το μέλλον της Ένωσης. Καταφέραμε να ενσωματώσουμε την ενεργειακή στρατηγική στις νομικές ε, πράξεις της Ένωσης. Συστάθηκε ο ειδικευμένο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τα Ενεργειακά Ζητήματα. Γίνονται δηλαδή ε, σημαντικά και αυτά βήματα για την ολοκλήρωση της ε, ενίας αγοράς. Τώρα, μπορούμε να επαναπαυθούμε στις δάφνες μας, αφήστατα όχι. Αυτό προκύπτει και από τη συζήτησή μας. Έχουμε τις οδηγίες, ε, ε, επειδή σας μιλούσα για τις νομικές πράξεις ε, προηγουμένως, έχουμε διάφορες οδηγίες, αλλά το σημαντικό είναι η εφαρμογή από πλευράς κρατούς μέλους της οδηγίας και επίσης η ρύθμιση των πρακτικών τεχνικών λεπτομεριών. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι αδυνατεί να δράσει από μόνο του και τα τελευταία χρόνια ε, σε συνεργασία με τον κύριο Ρόιλε και άλλα μέλη της Επιτροπής Βιομηχανίας ε, συμβάλαμε σε μεγάλο βαθμό στις συζητήσει που γίνονται για αυτό το ευρωπαϊκό επίτευγμα. Τώρα όμως φτάσαμε στην φάση εφαρμογής και άρα θα πρέπει να περάσει η σκητάλη στις κυβερνήσεις των κρατών μελών και τα εθνικά κοινοβούλια. Εξού και ιδιαίτερη σημασία της σημερινής διάσκεψης εφόσον ε, με την παρουσία των βουλευτών των Εθνικών Κοινοβουλίων ε, υπάρχει η δυνατότητα να συμβάλλουν και τα Εθνικά Κοινοβούλια στο ε, συνολικό αυτό εγχείρημα. Θα αντλούσα τα εξή ε, ε, συμπεράσματα από την ε, σημερινή συζήτηση. Οφείλουμε να εστιάσουμε την προσοχή μας στα θέματα εφαρμογής των οδηγιών και θα ήθελα να σταθώ λίγο στο ενεργειακό πακέτο. Υπολείπεται μεγάλο έργο αλλά μην ξεχνάτε ότι όσο καλή και αν είναι η νομοθετική ρύθμιση, δεν επαρκεί. Χρειαζόμαστε αγωγούς και καλές υποδομές και Η έμφαση που αποδώσαμε σε αυτά το ε, απόγευμα, σε ημερινή μας συζήτηση, νομίζω είναι αυτή η απόδειξη. Η ύπαρξη των υποδομών, η ποιότητα των υποδομών, η ποιότητα ε, των υπηρεσιών των ευφυών δικτύων πρέπει να κατοχυρωθούν. Θα ήθελα λοιπόν να συνοψίσω τα βασικά συμπεράσματα της συνεδρίας. Ως προς ενεργειακούς ε, διαδρόμους, και τις υποδομές. Προέκυψε σήμερα με σαφήνεια πως σημειώνονται βασικές διαφορές ε, ανάλογα με το κράτος μέλος ως προς την ενεργειακή διαφοροποίηση, αν θέλετε διαφοροποίηση του ενεργειακού εφοδιασμού. Η σύνθεση του ενεργειακού μείγματος, ο πετρέλαιο και φυσικό αέριο, διαφέρει σε μεγάλο βαθμό από τη μία χώρα στην άλλη. Οι βαλτικές χώρε ε, Φερρυπίν, εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από μία και μόνο ενεργειακή πηγή. Ε, οι χώρες κεντρικής Ευρώπης επίση κατά 80% εξαρτώνται από την ίδια πηγή, τη Ρωσία δηλαδή, και ταυτόχρονα οι Ιταλοί ε, συνάδελφοί μα συνέβαλαν σε μεγάλο βαθμό στην συζήτηση με τις παρεμβάσεις τους. Η Ιταλία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την Βόρεια Αφρική. Ε, ε, άρα η Ιταλία αν είχε τελικά πρόσβαση ε, στην Ρωσία, αυτό θα ενίσχυε την διαφοροποίηση της χώρας αυτής. Για την διαφοροποίηση των πηγών. Δεν εννοώ ότι θα πρέπει να εστιάσουμε σε ε, ε, μία, στην τάδε ή στη δίνα ενεργειακή πηγή. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι η διαφοροποίηση. Και θα ήθελα να σας δώσω και κάποια συγκεκριμένα παραδείγματα. Να μπούκο. Είναι προφανές ότι πρέπει να αναφερθώ κατά προτεραιότητα σε αυτό το πρόγραμμα. Είμαι προσωπικά πεπισμένος πως ο Ναμπούκο θα είναι ένας χρησιμότατος ενεργειακός διάδρομος ε, για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θα συμφωνήσω με αυτά που μας ε, είπε ο κύριος ε, Αράτσκι, υπάρχει καλύτερη λύση σε σχέση με το South Stream. Ε, ε, κατά πάσα πιθανότητα η ιδεατή λίστα ήταν συνδυασμό των δύο. Αλλά πραγματικά πέρα από, τους, από τις οδούς διανομής της ενέργειας πρέπει να αποδώσουμε το δέον βάρος στην διαφοροποίηση. Επίσης, ε, φυσικό αέριο από την Κασπία θάλασσα για να μην εξαρτώμαστε μόνο αποκλειστικά από την ε, Ρωσία. Οι τερματικοί σταθμοί του υγροποιημένου φυσικού αερίου επίσης έχουν ιδιαίτερη σημασία για την ενεργειακή διαφοροποίηση και συζητήθηκε με μακρόν το ζήτημα σήμερα. Ε, χάρη σε αυτό θα έχουμε καλύτερη ισορροπία ανάμεσα στην προσφορά και τη ζήτηση. μόλις ε, αρχίσουν να λειτουργούν οι εξωτερικές ε, υποδομές ε, θα πρέπει να ασχοληθούμε με την κοινή διαπραγματευτική μας θέση ενώπιον τρίτων χωρών. Είπαμε ήδη πως η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η πιο σημαντική αγορά 500 εκατομμύρια καταναλώτες έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό κανονικά πρέπει να λειτουργεί προ όφελό μας στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων. Μας δίνει πυγμή ισχύ, αν θέλετε, στη διαπραγματευτική αρένα. Για την Πολωνία, παραδείγματο χάρη, Ε, λειτουργήσε αισίως το σύστημα όταν διαπραγματευόταν διμερείς συμφωνίες προμήθειας φυσικού αερίου. Είναι προφανές πως η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πολλά να κερδίσει από την ε, υιοθέτηση μιας ε, κοινή ενιαίας προσέγγισης για τα ενεργειακά ζητήματα. Καλωσορίζω επίσης το ότι η Πολωνική Προεδρία θα ασχοληθεί επισταμένα με αυτό το θέμα και επικροτώ την, ενεργεια... την ιδέα της ενεργειακής αλληλεγγύης ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Είναι πραγματικά ζωτικό το ζήτημα. Για τις ε, εσωτερικές ε, υποδομές, 7 άτομα αναφέρθηκαν σε αυτό και πολύ σωστά ανέφεραν ότι χρειαζόμαστε ευέλικτα εγχώρια δίκτυα και όχι μόνο ενεργειακού διαδρόμους που θα μας συνδέουν με τρίτες χώρες. Ε, ε χρειάζεται να εξασφαλίσουμε ε, συνδεσιμότητα ε, ανά την επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είτε μιλάμε για το Βορρά, το Νότο, είτε την Ανατολή και τη Δύση Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χρειαζόμαστε μια πολυδιάστατη προσέγγιση που να καλύπτει όλη την επικράτεια της Ένωσης. Θα αρχίσουμε βεβαίως εφαρμόζοντας τους κανόνες που ήδη υπάρχουν και από εκεί και πέρα θα μπορέσουμε να αυξήσουμε την απόδοση ε, της ε, ε, υφιστάμενης δυναμικότητάς μας και, και χρειαζόμαστε φυσικά νέα δυναμικότητα καθώς και χώρους αποθήκευσης. Ένα δεύτερο στάδιο, αν ναι να πω ότι είναι αναπόφευκτο αυτές οι νέες ευρωπαϊκές επενδύσεις εφόσον επιθυμούμε να δημιουργήσουμε νέα δίκτυα. Ακούσαμε πολλοί άριθμα παραδείγματα ευέλτης πρακτικής συνεργασία ανάμεσα ε, σε δύο κράτη-μέλη, παραδείγματος χάρη και διασύνδεση των δικτύων τους. Αυτό βοηθάει τις ε, περιφέρειες, τις περιοχές της Ένωσης να μειώσουν την ενεργειακή τους εξάρτηση, αλλά αυτό δεν αρκεί. Χρειαζόμαστε ένα νομικό πλαίσιο, αλλά και μια αποτελεσματική αγορά, όπως είπε ο κύριος Αράτσκι. Ε, δεν είμαστε ανταγωνιστές ε, μέσα στην ενιαία αγορά. Συνεργάτες είμαστε και οφείλουμε να δείχνουμε αλληλεγγύη, όπως έλεγα προηγουμένως. Πάντως, ε, έχει σημειωθεί μια καμπή σε σχέση με το παρελθόν, σε σχέση, παραδείγματος με τη συνεδρία της 4ης Φεβρουαρίου, όπου το Συμβούλιο αποφάσισε να υποπειραθεί μέχρι το 2014 να έχει ολοκληρώσει αυτή την ενιαία αγορά με παράλληλη δέσμευση κατάργηση των ενεργειακών νησίδων μέχρι το 2050. Ε, προφανώς θα συναντήσουμε πολλά προσκόμματα στο δρόμο αυτό ως προς τις υποδομές και τη, τον τρόπο λειτουργίας εσωτερικής αγοράς. Θα ήθελα συγκεκριμένα να αναφερθώ σε δύο φραγμούς. Πρώτον το θέμα της αδειοδότησης. Είναι ένας από τους βασικότερους ε, είναι χρονοβόρες και εξαιρετικά περίπλοκες μέχρι στιγμής οι διαδικασίες αδειοδότησης και σε πολλές περιπτώσεις ε, χρειάζεται πάνω από 10 χρόνια για αδειοδότηση για συνοριακά προγράμματα. Παράδειγμα, στον 21ο αιώνα οφείλουμε να την επισπεύσουμε τη διαδικασία διοδότηση και ή δυνατόν να έχουμε και μία μονοαπευθυντική θηρίδα, όπω ε, ε, ονομάζεται, One Stop Shop, ένα ενιαίο σημείο επαφή για τη χορήγηση αδειών. Δεύτερο πρόβλημα, βασικότατο, έλλειψη πόρων. Χρηματοδότηση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί ότι μέχρι το 2020 πάνω από 200 δι ευρώ θα χρειαστούν για να διευρυνθούν, να επεκταθούν τα ευρωπαϊκά ενεργειακά δίκτυα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αρχίσαμε ήδη την συλλογή και την ε, εκπόνηση συμπιλημάτων με τα απαιτούμενα στατιστικά δεδομένα θα απαιτηθούν ε, σοβαρές επενδύσεις και για τον Αμπούκο και για το South Stream. Θεωρώ δε ότι έχουμε καθυστερήσει υπερβολικά για την εξέβρεση των απαιτούμενων πόρων και είναι ε, σίγουρο ότι θα πρέπει να επενδύσει και ο ιδιωτικός τομέας. Να μην τα αφήσουμε όλα στην αγορά. Χρειάζεται μια επένδυση ευρωπαϊκή ορισμένη, το είπαν. Ναι, όχι. Τόσες πολλές προτεραιότητες δεν είναι προτεραιότητες. Πρέπει να δούμε τι είναι σημαντικό να πραγματοποιηθεί και τι είναι λιγότερο ε, σημαντικό. Και αν κατορθώσουμε παρόλη την γραφειοκρατία να πραγματοποιήσουμε έργα και, τα και παρά τα προβλήματα χρηματοδότησης, θα είναι σημαντικό να έχουμε το καλό δίκτυο και θα χρειαστούμε ένα ευφυές δίκτυο. Ακούσαμε πολλά παραδείγματα προβλημάτων Ήδη ακούσαμε ότι θα είναι δυνατόν να πραγματοποιήσουμε 10% εξοικονόμηση ενέργειας απλώς με ένα καλό ενεργειακό δίκτυο, διότι αυτό θα επιτρέψει να, να μετακινήσουμε τη ζήτηση, να την μετατοπίσουμε αν το 2020 χρειαζόμαστε μια επένδυση 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων, μας λέει η Κομισιό, θα πρέπει να θυμηθούμε τα όσα λέχθηκαν. Μας χρειάζεται ένα ευφυές δίκτυο, αλλά αυτό απαιτεί επίσης μετρητές ευφυής, ούτως ώστε όλα να λειτουργούν καλά. Και αυτοί οι ευφυείς μετρητές επιτρέπουν να ευαισθητοποιήσουμε τους καταναλωτές στα νοικοκυριά και αυτό θα ήταν ένα πλεονέκτημα για μια κατανάλωση ενέργειας ε, πιο συνειδητής γενικά. Είναι σημαντικό να μην ξεχνούμε ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έλαβε μια απόφαση αποφασίστηκαν ε, κοινοί κανόνες, κοινά πρότυπα και μέχρι το 2020 στόχος είναι να μην έχουμε 10 αλλά 80% των κτηρίων που να είναι ε, εξοπλισμένα με ευφυείς μετρητές. Σχετικά με την στρατηγική θα ήθελα να κλείσω λέγοντας ότι μιλούμε ίσως περισσότερο για ασφάλεια εφοδιασμού από ότι ε, για τα άλλα θέματα όπως είναι η διατηρησιμότητα, η αηφορία. Δεν πρέπει όμως και αυτή να την ξεχνούμε, διότι είναι σημαντική. Από την άποψη αυτή θα ήθελα να αναφερθώ ε, στην ενεργειακή στρατηγική 2050 Πρόκειται για μια στρατηγική που προβλέπει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να είναι τελείως ανεξάρτηση από τον άνθρακα και από τα ορυκτά καύσιμα μέχρι το 2050 για την ώρα. Πρέπει να το εξετάσουμε το θέμα αυτό ήδη από τώρα αν θέλουμε να έχουμε αποτελέσματα το 2050. Λόγω των σημερινών συζητήσεων είναι σαφές ότι ε, σε περίπτωση, σε κατάσταση κρίσης όπως σήμερα, ο τομέας ο ενεργειακός αποτελεί μέρος του προβλήματος, αλλά να ακούσω τα όσα λέχθηκαν, δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι ο ενεργειακός τομέας είναι και μέρος ε, της λύσης και θα πρέπει όλοι μαζί να εργαστούμε προς τον σκοπό αυτό για το μέλλον. Ευχαριστώ κυρίες και κύριοι. Ο κύριος Ρόιλ άνοιξε τη συνεδρίαση και σε μένα ε, και σε μένα, εγώ πρέπει να κλείσω, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλα ε, τα μέλη Εθνικών Κοινοβουλίων, Ευρωκοινοβουλίου και την Ουγγρική Προεδρία που οργάνωσε εδώ αυτή την συνεδρίαση. Ευχαριστώ ε, όσους ήρθαν εδώ που συνέβαλαν και ευχαριστώ όσους εξέφρασαν εδώ τη γνώμη τους. Ευχαριστώ. Λύεται τη συνεδρία.